Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Πρώτα, έχουμε ψηφοφορία. Πρόκειται για το μέτωπο παγκοσμιοποίησης. Το πρώτο θέμα αφορά τη Γαλλικία το Wearing Apparel, Ισπανία. Και υπάρχει μια προσθήκη στην πρώτη παράγραφο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με 29 ψήφους κατά. Και υπάρχει και πρόταση της ΓΚΟΕ για μια νέα παράγραφο 3α υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προτείνεται και ένα παράγραφο στο 3β υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Και πάλι πρόταση γκουε, νέα παράγραφος 3 γάμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη επιστολή, υπέρ, κατά. Α, ηλεκτρονικά πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Ωραία, τότε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Εγκρίθηκε. 40 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Συνεχίζουμε και περνάμε στην νομοδότηση για την κινητοποίηση του Ταμείου για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Αφορά την Έριξον, είναι μια σουηδική πρόταση υπέρ. Πάλι ηλεκτρονικά, ναι, ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε γιατί πρόκειται για την επιστολή αυτή καθε αυτή. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 40 ψήφους υπέρ και μία κατά. Αυτό ήτανε από ψηφοφορίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα και να περάσουμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, ε, για να εξετάσουμε το σημείο 8 που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Εδώ καλωσορίζουμε την κυρία Τάισεν, την Επίτροπο Τάισεν, εδώ στην Επιτροπή μας. Θα μας παρουσιάσετε την πρόταση της Επιτροπής για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση, θα έχουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις από τους ευρωβουλευτές. Οπότε κύριε Τάισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε για να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω την πρότασή μας για οδηγία όσον αφορά διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας. Όπως ξέρετε, είναι ένα από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουμε στον κοινωνικό πυλώνα. Και απαντάει ουσιαστικά και στο έτοιμά σας να αντιμετωπίσουμε το θέμα των συνθηκών εργασίας υπό το φως της, ε, των νέων μορφών απασχόλησης που έχουν εμφανιστεί. Έχετε ήδη από πέρυσι εγκρίνει δύο ψηφίσματα, ένα για το κοινωνικό πυλώνα, τα κοινωνικά δικαιώματα, Ροντρίγκες, και ένα άλλο για τις συνθήκε εργασίες ε, και την, ε, τις επισφαλείς ε, μορφές εργασίας. Και, οι δύο, και τα δύο αυτά κείμενα ακριβώς αυτό ζητούν, να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες μορφές εργασίας. Θέλουμε λοιπόν ε, καλύτερες συνθήκε εργασίας με περισσότερη διαφάνεια και δικαιώματα είναι κάτι που τα πάντα στην καρδιά της Ευρώπης. Η κοινωνική διάσταση έτσι καλώς εξελίχθηκε με την ευάθυνση της Ευρώπης υπέρ και των επιχειρήσεων και υπέρ της ζωής εκατομμυρίων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτασε πια η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς αυτή την κατεύθυνση. Η δικιά μας η πρόταση εξυγχρονίζει τους υπάρχοντες τους κανόνες για τις ηθίκες εργασίας με ειδικό στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και εκείνοι που έχουν ε, μη ε, ε, τυπική εργασία, που έχουν άτυπες μορφές εργασίας, θα χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων που θα καθορίζονται με σαφήνεια. Η πρόταση αυτή λοιπόν πρώτα απ' όλα ε, ξυγχρονίζει τα δικαιώματα για τον κάθε εργαζόμενο. Και αυτό γίνεται βάσει μιας γραπτής δήλωσης η οποία θα υπάρχει. Δεύτερον, η πρόταση θέλει να προσαρμόσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο νέο κόσμο εργασίας έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να υποφελούνται από τα δικαιώματα αυτά. Οπότε θέλουμε να βάλουμε ένα κατώτατο όριο ε, δίκαιων συνθηκών ε, εργασίας με δικαιώματα για όλες τις μορφές εργασίας, για όλες τις συμβάσεις. Η πρόταση βέβαια δεν ε, λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν και άλλες νέες μορφές ακόμα εργασίες. Στόχος της πρότασης αυτής είναι να θέσει ένα πλαίσιο που, μέσα στο οποίο να μπορέσουν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερες διαφορετικές μορφές εργασίας ενδεχομένως στο μέλλον και να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τους νομοθέτες, για τα δικαστήρια και ισότιμες συνθήκες για όλους. Όπως γνωρίζετε, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σε δύο στάδια, ώστε να αναθεωρηθεί ενδεχομένως η οδηγία για τη γραπτή δήλωση. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα αυτή την πρόταση, κάτι το οποίο το ανέφερε και κατά τις διαβουλεύσεις. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία όσον αφορά ε, τον ε, σκοπό. Σε μια σύγχρονη και ελαστική αγορά εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι γραπτός για τις βασικές συνθήκες της εργασιακής τους αυτής σχέσης. Υπό τους σημερινούς κανόνες, οι χώρες μέλη μπορούν να αποφασίσουν ποιες, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι καλύπτονται από μια τέτοια διάταξη. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που είναι εκτός. Εκείνοι που εργάζονται περιστασιακά ή με συμβάσει ε, διαλήψης απασχόλησης, πλατφόρμα. Για κάποιους εργαζόμενους όμως αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται κάτω από επισφαλείς συνθήκες. Δικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε τη δυνατότητα αποκλεισμού εργαζόμενων από την κάλυψη της οδηγίας και συνεπώς ο σκοπός αυτός της οδηγίας να ανταποκριθεί στην έννοια των εργαζόμενων έτσι όπως αναφέρεται ε, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όλοι οι εργαζόμενοι που για ένα διάστημα προσφέρουν υπηρεσίες για κάποιον, υπό κάποιου, επίσης οπότε λαμβάνει και κάποια ανταμοιβή για την υπηρεσία του αυτή, θεωρείται εργαζόμενος. Όταν μιλάμε λοιπόν τώρα για έναν ενιαίο ορισμό για το τι είναι εργαζόμενος, σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κάποιες κατηγορίες και δεν μένει κανένας απ' έξω. Με την οδηγία αυτή λοιπόν θα υπάρξει ένα επιπλέον εργαλείο για να είμαστε σε θέση να ξέρουμε κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί καλύπτονται. Όντως, δηλαδή, εφόσον εμπίπτουν στο εύρο εφαρμογή τη οδηγία, κατά πόσο όντως γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ε, εργαζόμενους που θα καλύπτονται επιπλέον από αυτή τη ρύθμιση. Δεύτερον, η πρόταση αυτή εξυγχρονίζει και το τι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στον ε, εργαζόμενο. Επιπλέον από τις σημερινές ε, πληροφορίες θα υπάρχουν και παραπάνω που θα μιλούν για το χρόνο και θα δίνουν και συγκεκριμένες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα και τις ώρες εργασίας. Επίσης θα μιλάνε πληροφορίες αυτές και για την κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον οι απαιτήσει ε, αυτές θα πρέπει να δίνονται στον εργαζόμενο από την πρώτη ημέρα εργασίας του και όχι σε δύο μήνες όπως λέει το σημερινό κείμενο. Και αυτό για να αποφεύγεται η αδήλωτη εργασία. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει και κάποια επιπλέον ουσιαστικά δικαιώματα στην πρόταση που έχουν να κάνουν με το στόχο του να προσφέρουμε κάποια ελάχιστη προβλεψιμότητα στους εργαζόμενους και να υπάρχει επίσης ε, ε, ευελιξία χωρίς όμως να υπάρχει αβεβαιότητα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει ε, στο κείμενο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα για τη δοκιμαστική περίοδο. Λέει ότι η δοκιμαστική περίοδος πρέπει να περιορίζεται σε 6 μήνες. Εκτός αν ρητά δικαιολογείται μια άλλη περίοδος, αν έχει θέση ε, managerial, ας πούμε, ο εργαζόμενος. Η αρχή 5 το λέει ότι πρέπει η δοκιμαστική περίοδος να έχει εύλογη διάρκεια. Δεύτερον, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα παράλληλη απασχόληση, να μπορεί να δουλέψει δηλαδή και για άλλον εργοδότη ο εργαζόμενο. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η ρήτρα αποκλειστική απασχόληση και περιορισμό που να λέει ότι είναι ασύμβατο ο εργαζόμενο να έχει και μια άλλη δουλειά. Εμεί πιστεύουμε ότι κανένα εργαζόμενο δεν θα πρέπει να προσφέρει κατά αποκλειστικότητα την εργασία του σε κάποιον εργοδότη. Εκτός βέβαια από μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν υπάρχουν ρήτρες ασυμβατότητας, αλλά τότε θα πρέπει να δικαιολογείται αυτό από θεμητούς λόγους όπως είναι η προστασία του επιχειρηματικού απορρίτου ή η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Και πάνω σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Συμβάσει μηδέν ωρών με αποκλειστικότητα σε ρήτρες δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη. Και τρίτον, ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να ξέρει από πριν πότε θα πρέπει να δουλέψει. Οπότε να μπορεί, αν θέλει, να δουλέψει και κάπου αλλού ή να ασχοληθεί με την οικογένειά του, αν θέλει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που δουλεύουν με βάρδιες, που τις καθορίζουν οι εργοδότες. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για υπερορίες που μπορεί να συμβούν περιστασιακά μέσα στη χρονιά. Όχι. Λέμε ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να έχει το δικαίωμα όποτε θέλει να φωνάσει τον εργαζόμενο να εργαστεί. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξέρουν ποια, ποια είναι τα ωράρια αναφοράς βάσει των οποίων ε, θα κληθούν να εργαστούν και θα πρέπει έγκαιρα πριν να το γνωρίζουν εάν υπάρξει κάποια αλλαγή. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα προβλέπεται για μια πιο σταθερή απασχόληση και υπάρχει υποχρέωση για γραπτή απάντηση. Σίγουρα ε, πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία, όμως υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να παγιδεύονται σε συμβάσεις που δεν δίνουν καμία βεβαιότητα και που δεν επιτρέπουν και καμία αλλαγή σε πιο μόνιμη απασχόληση. Από το διάλογο φάνηκε ότι εμεί προτείναμε πως οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν περισσότερη βεβαιότητα στις συμβάσεις τους και να έχουν γραπτή απάντηση από τον εργοδότη που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και του εργοδότη και του εργαζόμενου. Έπειτα, το δικαίωμα σε δωρεάν κατάρτιση. Οι εργοδότες πρέπει και βάσει των συλλογικών συμβάσεων να προσφέρουν κατάρτιση στους εργαζόμενους. Και είναι πολύ σημαντικό η κατάρτιση αυτή να, προστατε... να προσφέρεται χωρίς διακρίσεις σε βάρος αυτών που έχουν άτυπες μορφές απασχόλησης. Και το κόστος δεν πρέπει να το επομίζεται ο εργαζόμενος. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα δικαιώματα θα προσφέρονται όντως, προτείνονται και οι μορφές εφαρμογές του στο κοινωνικό κεκτημένο, για παράδειγμα, με δικητικές διαδικασίες, οι ποινές, με επανόρθωση κλπ. Για να ολοκληρώσω, στόχος μας είναι να προσφέρουμε κάποιες ελάχιστες ε, δίκαιε ηθίκες εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη για όλου του εργαζόμενους με όποια μορφή και αν απασχολούνται. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο και ελπίζω να βοηθήσετε κι εσείς να προχωρήσει η, τροπολογία, η, συγγνώμη, η πρόταση αυτή στα πλαίσια τη σημερινή μα θητεία. Το Συμβούλιο έχει ήδη αρχίσει να συζητάει την πρόταση αυτή και σίγουρα ε, μέχρι το τέλος της Βουλγαρικής Προεδρίας θα έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα λέω ότι όπω πάντα είμαστε και τώρα έτοιμοι να βοηθήσουμε του συνομοθέτε για να ε, καταλήξουν σε απόφαση πριν από τα τέλη της χρονιάς. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. κύρια Πρόεδρε, συνηθίζουμε να λέμε chairman, αλλά chair θα έπρεπε να πω εδώ. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα προς τους πολίτες μας και προς τον κόσμο. Ότι δηλαδή στην Ευρώπη είμαστε ενωμένοι να υποστηρίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε για να προσθέσουμε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ αυτό κοινωνικών δικαιωμάτων και να προωθήσουμε την ε, κοινή μας ε, θέση για σήμερα και για το μέλλον υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ και είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τάισεν για την εισαγωγή που μας κάνατε. Θα περάσουμε απευθείας ε, στους συντονιστές που μπορούν ε, να θέσουν τα ερωτήματά τους. Ε, Ντάβιτ Κάζα πρώτος. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Και προσπαθήστε να μην μακρηγορήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την παρουσίαση που μας κάνατε. Η οδηγία θα επιβάλλει ε, και όρους εργασίας για τις νέες μορφές ε, συμβάσεων. Αλλά ε, πολλοί επιλέγουν ε, τις ελαστικές μορφές εργασίας ε, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Είναι η μόνη ευκαιρία εργασίας που έχουν. Μήπως έτσι καταστρέψουμε όμως αυτή τη δυνατότητα, εννοώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε η οδηγία αυτή να μην δημιουργήσει προβλήματα και σε αυτή τη μορφή εργασίας στην αγορά εργασίας. Χαβιέ Λόπες ο επόμενος ε, στη θέση του, της κυρίας Ιονκερίους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα η ομάδα μας θα ήθελε να ε, πει ότι καλωσορίζει ιδιαίτερο στην πρωτοβουλία της Επιτρόπου θεωρούμε ότι πρόκειται για πάρα πολύ ε, σοβαρή και σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την ευκαιρία ε, μέσω αυτού του κειμένου να ε, βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και κυρίως να καταπολεμήσουμε την αβεβαιότητα. και πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί αλλάζουν τα πράγματα στην κοινωνία και πρέπει και εμείς ε, να προσαρμοστούμε. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό ε, κοινή βάση δικαιωμάτων και προϋποθέσεων και όρων, ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη κοινή μάζα προτύπων, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και εμείς να ανακτήσουμε την ε, νομοποίηση που πρέπει να έχουμε στα μάτια των πολιτών μας και βεβαίως μετά από τον κοινωνικό πυλώνα θα έχουμε άλλο ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα από την πλευρά της Κομισιόν. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Εξάλλου είμαστε βέβαιοι ότι με αυτήν την πρωτοβουλία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις νέες τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας. Και εξηγούμε. Γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η ανάκαμψη, αλλά ε, επειδή έχει αλλάξει η αγορά εργασίας δεν δημιουργούνται ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή έχουμε όλο και πιο ευάλωτους εργαζόμενους βλέπουμε και την οικονομία ε, η οποία λειτουργεί βάσει αυτών των πλατφορμών με αβέβαιες συνθήκες εργασίας. Βλέπουμε πολλές νέες τάσεις στην αγορά εργασίας ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι τούτη εδώ η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτοί οι νεοτερισμοί ε, της ε, αγοράς εργασίας, ε, κυρίως τις άτυπες μορφές, όπως είπε και η ίδια η Επίτροπος. Τρίτο σημείο. Η ομάδα μας έχει δεσμευτεί όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα και όσον αφορά ε, έναν ικανό βαθμό προβλεψιμότητας ε, ε, των, της εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Είναι πάρα πολύ θετικό που συνεργαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μακιντάιερ, όχι δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ η κυρία Μακιντάιερ. Θα πάρετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να συμφωνήσω με το ερώτημα του κυρίου Κάζα, εάν η οδηγία αυτή δεν θα επιφέρει περιορισμό της ευελιξίας και μήπως θα υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες για μαύρη παράνομη εργασία και έτσι να μην πετύχουμε τον στόχο μας που είναι περισσότερη βεβαιότητα για τους εργαζομένους. Αντιθέτως, ε, μήπως δούμε περισσότερα εμπόδια και ε, τρόπους παράκαμψης των κανόνων. Ευχαριστώ. Then we go to, ε, Mr. Περνάμε τώρα στον κύριο Καλβέ Σαμό, που είναι και εισηγητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Καθότι γνωρίζω ότι κατέχετε πολύ καλά την γλώσσα του Μολιέρου. Λοιπόν, Ε, εδώ τώρα μπήκατε λίγο στα δικά μου τα χωράφια και σας λέω ότι εγώ είμαι εισηγητής ε, του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν ε, το ακούτε με ευχαρίστηση. Σας το λέω για να είστε προετοιμασμένοι ότι θα με βλέπετε μπροστά σας συχνά γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός καθότι ο ρόλος μου είναι λίγο να συνδέσω τις θέσεις και τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα. Αλλά ε, παρόλα αυτά πιστεύω ότι εδώ κάνουμε ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό το οποίο μπορεί να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ελκυστική μονάχα εάν είναι και κοινωνική και εάν την εκλαμβάνουν ως κοινωνική Ευρώπη οι πολίτες της. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν και χαίρομαι γι' αυτό. Οι αρχές τις οποίες εξαγγείλατε, κατά την άποψή μου και με κάποιες μικρές διαφορές, με βρίσκουν σύμφωνο και εν πάση περιπτώσει θεωρώ τις αρχές που εξαγγείλατε αποδεκτές. Μετά βέβαια θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, τις δυσκολίες υλοποίησης, τις δυσκολίες εφαρμογής ε, γιατί όπως είπατε και εσείς η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και αυτό οφείλεται σε πολλαπλά αίτια. Μπορεί οι δομές να είναι διαφορετικές, οι συνήθειες παραδόσεις διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει απλά να δούμε ποια είναι ε, τα οριζόντια ελάχιστα ελάχιστα δικαιώματα. Πράγμα εκ των ουκάνευ για το ε, κοινωνικό ε, πρόσωπο που θέλουμε να έχουμε. Μιλάγαμε σήμερα το πρωί με τον επικεφαλής της Eurofound και ακριβώς αυτό το ίδιο συζητούσαμε. γιατί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ένα δικό μας ε, πρόσημο το οποίο θα μας διαφοροποιεί από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ε, ε, αυτό το κείμενο είναι πολλαπλό αλλά ιδιαιτέρως και αυτή η δράση παρουσιάζει το εξειδικευμένο ενδιαφέρον το οποίο πώς να σας το εκφράσω Εάν ήθελα να είμαι ε, αισιόδοξο, θα έλεγα ότι είναι το έμβριο, αν όχι το προέμβριο, ε, της ε, κοινωνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά πολλά θέματα, υποχρεωτική κατάρτιση, ε, ε, καθορισμός ελαχίστων ορίων και για πολλά άλλα οπωσδήποτε θα πρέπει να ακούσουμε τους πάντες, ε, όλους τους εμπλεκόμενους, εργοδοσία, εργαζόμενους, συνδικάτα και η εργοδοσία είναι μοιρασμένη, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες. Και εμείς από την δικιά μας πλευρά λέμε ότι θα παραμείνουμε ε, στις θέσεις που εκφράζω σε αυτό το μικρό βιβλίο που σας ε, ε, προσέφερα και όπου αναφέρει την, τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης στον 21ο αιώνα. Vous, en, vous me le faites. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι εμείς η δουλειά μας είναι να κάνουμε ένα υλοποιήσιμο μοντέλο και για να είναι υλοποιήσιμο θα πρέπει καλά και σωστά να προβλέψουμε και να μετρήσουμε τα κόστη βράχη, μέσο και πρόθεσμα. Και επίσης απαραίτητο συστατικό και στοιχείο είναι και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αλλά γενικώ έχω ένα πολύ καλό επικοδομητικό πνεύμα και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και οι ιδέες εκ πρώτης όψεως φαίνονται σωστές και τώρα ας ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπη. Thank you. Then... <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Περνάμε στην QNGL. Ειρήνα ρόνια παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε και ευχαριστώ που ήρθατε να μας παρουσιάσετε την πρότασή σας εδώ σήμερα. Η ομάδα μας εσημερίζεται τον στόχο να έχουμε μια ασφαλή αγορά εργασίας, ή εργαζόμενοι να γνωρίζουν ε, τις συνθήκες απασχόλησής τους και να υπάρχει ασφάλεια ως προς αυτές. Χρειαζόμαστε ισχυρές ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, που να διαπραγματεύονται τις συνθήκες με τους εργοδότες σχετικά με την κατανομή της εργασίας. Και γι' αυτό ως πολιτικοί, θα πρέ... ως νομοθέτες θα πρέπει να προσέξουμε πολύ εάν θέλουμε να επέμβουμε ε, στις συλλογικές συμβάσεις, διότι αυτές είναι ο πυρήνας σε μια ασφαλή αγορά εργασίας. Ο χρόνος εργασίας ε, είναι ένα θέμα το οποίο συχνά ε, διαπραγματεύονται οι ε, συλλογικές συμβάσεις. Χρειάζεται λοιπόν ασφάλεια για τον εργαζόμενο και χρειάζεται και η ευελιξία που θέλει ο εργοδότης. Και γι' αυτό ακριβώς ε, οι κοινωνικοί εταίροι συνήθως ε, ε, διαπραγματεύονται τα θέματα αυτά. Η πρόταση οδηγία αυτή παρεμβαίνει όμω σε αυτό και διάφορε συνδικαλιστικέ οργανώσει στην Ευρώπη ήδη το έχουν επικρίνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώ απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι επικρίσει αυτέ, ότι ανακατεύεστε στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. και συμφωνείτε με τον ισχυρισμό ότι η πρόταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε, τελικά σε απόφαση ε, του δικαστηρίου, ε, δηλαδή το, ένα, το, δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μπορεί να ακυρώσει η συλλογική σύμβαση με βάση αυτήν την οδηγία, αυτό θα ήταν ε, μάλλον κάτι πολύ ριζικό για την αγορά εργασίας μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στανόκα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ομάδα μας ε, γενικά επικροτεί τη νέα πρόταση που αποτελεί ένα βήμα ε, στην πραγματοποίηση των στόχων του κοινωνικού πυλώνα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι επικεντρώνεται στους εργαζομένους και ότι παρέχει βάση για καλύτερες συνθήκες εργασίες για τους εργαζομένους ε, ιδιαίτερα σε νέες μορφές θέσεων απασχόλησης ε, επισφαλής, σε, θέσεις, σε επισφαλής θέσεις Ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Καταρχάς, η οδηγία αυτή δεν αναφέρεται στους ασκούμενους. Αυτοί καλύπτονται μόνο από συστάσεις του Συμβουλίου. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες από πλευράς της ομάδας μας. Επίσης, θα θέλαμε πιο συγκεκριμένο κείμενο όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης, το δικαίωμα προσφυγής. Κατά τη γνώμη μας, οι διατάξεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ γενικές και θολές. Πιστεύουμε επίσης ότι χρειάζονται διευκρινήσεις σε σχετικά με το πότε και πώς θα παρέχονται πληροφορίες στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Αυτό είναι και ερώτηση, διότι το κείμενο δεν απαντάει στο ερώτημα αυτό. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ή κατά την υπογραφή της σύμβασης θα παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. Άλλη ερώτηση, πώς θα γίνεται αυτό. θα αρκεί η σύμβαση αυτή καθ' αυτή ή θα συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες σε μια σχετική σειρά κανόνων. Στη σύμβαση δηλαδή ή θα είναι ξεχωριστοί κανόνες. Και η σύμβαση αυτή θα προβλέπει και πιθανή απόσπαση του εργαζόμενου. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο, δεν είναι όμως αρκετά σαφές ότι θα πρέπει να ενημερώνεται ο εργαζόμενος ότι στο πλαίσιο της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει απόσπαση. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Ιδιαίτερα όταν ε, χρειάζονται οι εργαζόμενοι ε, συνδρομή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και εδώ θα θέλαμε να υποβάλουμε τροπολογίες, θα θέλαμε όμως να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Λάουρα Ατζέα τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την ε, Επίτροπο για αυτήν την ε, πρώτη γεύση που μας έδωσε και την εργασία που μας περιμένει. Ε, η βάση, ε, η πρόταση στη βάση της ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Θα πρέπει βέβαια να προσπαθήσουμε ε, μέσα από συνεργασία να προχωρήσουμε σε πραγματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Προβληματίζομαι λίγο και ίσως θα μπορούσε η Επίτροπος να αναφερθεί λίγο περισσότερο σε κάποια θέματα. Το ε, κόστος ε, για τις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες και πολύ μικρές. Το κόστος λοιπόν ποιο θα είναι ε, το δημοσιονομικό διορθώνω, το γραφειοκρατικό άχθος θα βαρύνει ε, τις ε, μικρές επιχειρήσεις στη στιγμή της εφαρμογής υλοποίησης οδηγίας. Επίσης, για τους εργαζόμενους που δεν υπόκεινται σε συλλογική σύμβαση, πώς θα εφαρμοστεί για αυτούς η οδηγία και κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις και ε, για τις εργασίες και τους εργαζόμενους που δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Ε, ας πούμε άσκηση, στάζ, κατηγορίες ε, εργασίας γενικώ που δεν καλύπτονται διότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η εκμετάλλευση ε, στα πλαίσια των ε, περιόδων μαθητείας, ε, στάζ, άσκησης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποιες εγγύσεις και όσον αφορά αυτά τα θέματα γιατί αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Και κάτι άλλο σε σχέση με τους αυτόνομους εργαζόμενους και το, το αφημί τους ε, εντάσσονται γενικά στην οδηγία αλλά σε περιπτώσεις όπου η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει ε, κάποιες ε, ειδικέ συνθήκες και κάποια ειδική προστασία για τους εργαζόμενους αυτούς με ποιο τρόπο η οδηγία μπορεί να τους καλύψει και επίσης με ποιο τρόπο θα μπορούσε ενδεχομένως να υλοποιηθεί διαφορετικά έτσι ώστε αυτή στην Ελλάδα τους λέμε εργαζόμενους με μπλοκάκι να μπορούν να καλυφθούν και από αυτήν την οδηγία. Ευχαριστώ. Then it's Mr. Martin. Ο κ. Μαλτάιν τώρα. Μάρτα. Όχι. Εγώ θα πάρω το λόγο, κύριε Μίλα. Ε, ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε που μας παρουσιάσατε την πρόταση αυτή που έχουν να κάνουν με, τις, με τη διαφάνεια στις συνθήκες εργασίας. Είναι κάτι πολύ σοβαρό βέβαια και θα αλλάξει τα δικαιώματα και των εργαζομένων και των εργοδοτών σε εθνικό επίπεδο. Από τα δικιά μας την πλευρά ε, πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός αυτός φαίνεται ότι είναι άκαμπτος, πολύ βαρύς, που αλλάζει πάρα πολλές συνήθειες και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι συμφωνούν οι εργοδότες οι μηχανισμοί μάλιστα αυτοί μπορεί να είναι και ξεπερασμένοι ή να είναι ξεπερασμένοι πολύ σύντομα δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οπότε τα συμφέροντα των εργοζομένων ποια είναι. Σίγουρα να έχουν ένα ευχάριστο χώρο εργασίας, αλλά δικαίωμά τους είναι και εργασία. Και όταν βλέπουμε τα κοινωνικά του 2017 διαπιστώνουμε ότι ε, μπορεί να υπάρχει ανάκαμψη στην Ευρώπη, Ευτυχώ, 10 χρόνια μετά την κρίση καιρό ήταν. Η ανάκαμψη αυτή όμω είναι πάρα πολύ δειλή και πολύ λιγότερη από ό,τι έχουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Και αν κοιτάξουμε ποιε είναι οι διάφορε παράμετροι απασχόληση, ε, ε, αγοραστική δύναμη των χωρών της Ευρωζώνης, η ομάδα μας πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να ελαφρύνουμε από διάφορες οδηγίες που βαραίνουν τους εργοδότες αντί να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση η οποία θα ε, κάνει περισσότερες καταστροφές από ό,τι νομίζουμε. Όπως και όλες οι διατάξεις που παίρνουμε εδώ και 50 χρόνια, ούτε και από αυτήν θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Η κυρία Γιουγκέριος τώρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγω ότι την ευχαριστώ που παίζει και το ρόλο του ακτιβιστή. Μ' αρέσει αυτό. Το λέω θετικά. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τον ορισμό του εργαζόμενου. Γιατί λέει ότι σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο για ένα χρονικό διάστημα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάποιον άλλον και ανταμείβεται για τις υπηρεσίες αυτές από τον κάποιο άλλο. Υπάρχουν νέες μορφές εργασίες, υπάρχει η πλατφόρμα για παράδειγμα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα οδηγία. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα γιατί αυτή η εργαζόμενη πλατφόρμα είναι πιο αυτόνομη. Και ρωτάω, θα καλύπτονται ή δεν θα καλύπτονται από αυτό τον ορισμό. Γιατί ένας εργαζόμενος πλατφόρμας κάνει αυτόνομα την εργασία του και δεν δουλεύει υπό κάποιον άλλον, τότε ανταποκρίνεται σε αυτόν τον κανονισμό ή μήπως αυτός ο ορισμός αποκλείει τους εργαζόμενους πλατφόρμας. Και το δεύτερο μου θέμα έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θα παίρνει ο εργαζόμενος. Και είπατε ότι πρόκειται για ελάχιστε προδιαγραφές. Η οδηγία επίσης στο άρθρο 19 μιλάει για πιο ευνοϊκές συνθήκες. Θα είναι ξεκάθαρο στην πρόταση ότι πρόκειται για ελάχιστες προδιαγραφές και ότι σε εθνικό επίπεδο το κάθε κράτος μέλος μπορεί να έχει έναν μεγαλύτερο κατάλογο απαιτήσεων όσον αφορά την πληροφόρηση που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη του. Τώρα θα πάρω εγώ το λόγο, λέει η Πρόεδρος, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και θα τα πω μα δεν μπορώ να δεχτώ την πρόταση αυτή ως έχει. Οι κοινωνικοί εταίροι στη Σουηδία και από τις δύο πλευρές, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μου, δεν είναι υπέρ της πρότασης αυτής. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, μεν, αλλά να, είναι πολύ προβληματικό να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ορισμό για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Αυτό έχει να κάνει με το σύστημα ε, συλλογικών ε, συμβάσεων και διαπραγματεύσεων. Στην χώρα μου θέλουμε ορισμούς που να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στις ε, ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας. Επίσης, κινδυνεύει να πλήξει και νομοθεσία στο τομέα το φορολογικό που είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα που δίνω. Θα μπορούσα επίσης να προσθέσω ότι εκφράζονται φόβοι από τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόμματα για το ότι ο κοινωνικός πυλώνας αποτελεί ένα κατάλογο γενικών αρχών που όμως αμφισβητούνται στα πλαίσια αυτής της πρότασης. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ενταχθούν σε όλα τα μοντέλα εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Και ότι πρόκειται για απειλή στην ίδια την επικουρικότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτές οι γενικές αρχές είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν στο εθνικό επίπεδο. Αλλά η αναθεώρηση αυτή της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση προκαλεί σύγχυση. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξανασκεφτεί και να επικεντρωθεί στη στήριξη των κοινωνικών εταίρων. Είναι πολλή δουλειά, μεγάλες οι προσδοκίες για το τι μπορούμε να πετύχουμε με τον κοινωνικό πυλώνα. Η αντίδραση όμως στη χώρα μου σήμερα είναι ότι θα έπρεπε να είναι κάτι πάνω στο οποίο θα συνεργαστούμε όλοι για να καταλήξουμε στην ίδια κατεύθυνση όλοι και όχι να πάει ο καθένας στη διαφορετική πλευρά. Δεν πρέπει να γεμίσουμε τον κοινωνικό πυλώνα με προτάσεις, με πράγματα γενικά, τα οποία στη συνέχεια δεν θα υλοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να υπερψηφίσω. Η Σουηδία τουλάχιστον δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει ούτε στο Συμβούλιο. Ήθελα να το υπογραμμίσω να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε μια πρόταση την οποία να μπορούν όλοι να υποστηρίξουν. Λέει πρόεδρος ε, Σαντέρ τώρα. Ε, η κυρία Σαντέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων επί της ε, προτάσεώς σας αναθεώρησης της οδηγίας ε, για πιο διαφανείς ε, και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Ως σκιώδης εισηγήτρια για την συνεταιριστική οικονομία ε, είχα την ευκαιρία να εργαστώ κυρίως για τις νέες μορφές εργασίας που τώρα αναδύονται καθώς επίσης και να μελετήσω το κατά πόσον πρέπει ή δεν πρέπει να πλαισιωθούν καλύτερα αυτά, αυτές τις νέες μορφές εργασίας. Κατά την έννοια αυτή λοιπόν προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Ακούσαμε ήδη μερικά. Ε, και εγώ έχω από τη σειρά μου, από τη μεριά μου κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω κύριε Επίτροπε. Ο ορισμός εργαζόμενου είναι ένας ευρύς ε, ορισμός ο προτινόμενος ε, γιατί ε, συμπεριλαμβάνει και κάποιους εργαζόμενους που τώρα θεωρούνται ε, ανεξάρτητοι. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ε, κάτι παραπάνω όσον αφορά αυτήν την κατηγορία των ανεξάρτητων ελεύθερων επαγγελματιών που μπαίνουν πλέον στον ορισμό. Επίσης, σε σχέση με άλλες οδηγίες, η ο ορισμός εργαζόμενων και εργοδοτών θα μεταφερθούν και επομένως θα εφαρμοστούν και στα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών οδηγιών ε, κυρίως ε, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες και εδώ έχω κάποια σχόλια, ίδια με αυτά που έκαναν προηγούμενοι συνάδελφοι Έχετε κάνει κάποιο προγραμματισμό, κάποιο σχεδιασμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχετε κάνει κάποιους υπολογισμούς. γιατί εάν δημιουργηθούν προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τότε θα έχουμε ακριβώς το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή να βελτιώσουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάμ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Αγαπητή Μαριάνε. βρίσκω πολύ καλό το ότι έχουμε την πρωτοβουλία αυτή και ότι ε, οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να αποτελούν κίνητρο, μπορεί να οδηγούν σε αντιδράσεις. Ε, εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτή η διαβούλευση σε δύο φάσεις με τους ε, κοινωνικούς τέρους Ε, δείχνουν ότι όσον αφορά τους στόχους συμφωνούμε, όχι όμως όσον αφορά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Και πού οφείλεται αυτό. Έχουμε ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δεύτερον, ε, ναι, φυσικά θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά αυτό σημαίνει ότι και όποιος πάει να δουλέψει κάπου να έχει κάτι στο χέρι του και μάλιστα γραπτός, ε, όχι μόνο προφορικά. Δεν αρκεί να του το εξηγήσουμε καλά, πρέπει να έχει ένα αποδεικτικό έγγραφο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Και κατόπιν φτάνω στους ε, έξι μήνες ε, της δοκιμαστικής περίοδου. Είναι σημαντικό αυτό, διότι μετά από τρεις μήνες δεν έχει κανείς απαραίτητα καθαρή εικόνα. Προτείνατε όμως να υπάρχουν και δυνατότητες παρέκκλησης. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι μορφή θα έχουν οι παρεκκλήσεις αυτές. Και τέλος, βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό όλοι να έχουν σαφή ορισμό του εργαζομένου. Γιατί, διότι έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις ε, δήθεν ξεκάθαρες, οι οποίες όμως υπονομεύονται από όλους τους διάφορους ε, κανόνες διότι υποτίθεται ότι υπάρχει ασφάλεια αλλά τελικά όλο και κάποιοι άλλοι κανόνες υπάρχουν λέει ο άλλος ότι εγώ είμαι αυτοπασχολούμενος ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα Ευχαριστώ Ευχαριστώ η Μαρία Χωαροντρίγες Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε Καλωσορίζω την Επίτροπο, χαιρετίζω και την πρόταση σχετικά με αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Νομίζω ότι αποτελεί πολύ καλό βήμα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαϊκός αυτός πυλώνας αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, δυνατόν να καταλήξουμε σε μια διακήρυξη σε πολύ ψηλό επίπεδο λόγω της πολύ καλής συνεργασίας Κοινοβουλίου και Επιτροπής και τελικά και του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στο Γκέτεμποργκ το Κοινοβούλιο είχε πολύ ισχυρή αντιπροσωπεία και αυτό ήταν πολύ σημαντικός πολιτικός παράγοντας. Εκπρόσωποι όλων των ομάδων που στήριξαν στην έκθεση του Κοινοβουλίου συμμετείχαν και έτσι εξασφαλίσαμε και την πολύ ευρία πλειοψηφία ε, υπέρ της πρότασης στο Κοινοβούλιο. Τώρα γνωρίζουμε ότι είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες του κοινού όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα και νομίζω ότι και πάλι θα χρειαστεί καλή συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θεωρώ καλή την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό αυτό που διακυβεύεται. Βλέπουμε νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, νέες, νέα είδη απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε όποια και να είναι η μορφή της απασχόλησης θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις για όλους τους εργαζομένους. Ε, σαφείς ε, συμβάσεις εργασίας πρώτον και δεύτερον πρόσβαση στην ε, κοινωνική προστασία. Γι' αυτό έχω ερώτηση προς την Επίτροπο. Ποια είναι η σχέση αυτής της οδηγίας με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Διότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο καλούνται οι υπογράφοντες της διακήρυξης ε, να δηλώσουν ποιο είναι το σύστημα κοινωνικής προστασίας ε, που να καλύπτει κάθε συγκεκριμένο εργαζόμενο. Φαίνεται σαν να είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ σημαντική και πολύ θετική, διότι έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ο κάθε εργαζόμενος να έχει πρόσβαση σε σύστημα κοινωνικής προστασίας ε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την λεπτομέρεια αυτή. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώς βλέπετε τη σχέση ανάμεσα σε αυτήν την οδηγία και στα όσα ετοιμάζετε για την κοινωνική προστασία. Μήπως μπορείτε να το αναπτύξετε λίγο αυτό. Τελική παρατήρηση για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Ας είμαστε δίκαιοι Προτού απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως είναι και σωστό. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε μέχρι την επίτευξη πιθανής συμφωνίας. Τελικά δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό η Επιτροπή αναθεωρεί την οδηγία οι κοινωνικοί εταίροι τώρα θα πρέπει να επανεξετάσουν το θέμα και εάν καταλήξουμε πάλι αυτή τη βδομάδα σε συμφωνία πάνω στην οδηγία αυτή όπως ελπίζουμε θα πρέπει πάλι οι κοινωνικοί εταίροι να ασχοληθούν με αυτήν. Με κανέναν τρόπο δεν υπονομεύει το κοινοβούλιο το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό. Φυσικά, δέχομαι τη δήλωση της Προέδρου που μίλησε ε, ως εκπρόσωπος της Σουηδικής Αντιπροσωπείας. Καταλαβαίνω την προοπτική της Σουηδικής πλευράς. Ωστόσο, η ομάδα S&D θα ε, στηρίξει την ιδέα αναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν πολύ σαφής ότι μίλησα με αυτή μου την ιδιότητα και δεν είμαι και βέβαιη ότι πρόκειται για αποκλειστικά σουηδική θέση. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε κάθε πρόταση της Σουηδίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, ε, της Ολλανδίας για παράδειγμα. Και δουλειά της κυρίας Τάισεν είναι να προσπαθήσει να συνδυάσει και να ικανοποιήσει όλες αυτές τις θέσεις. Κυρία Μπλίνκεβιτσούτε, σας παρακαλώ να να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση αυτή. Είμαστε ενθουσιώδεις όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα. Και αυτός ο κοινωνικός πυλώνας θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν ε, μπορεί να βοηθηθεί από διάφορα εργαλεία. Όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας για τις ελάχιστες συνθήκες εργασίας, και τι συμβάσει με όποια μορφή εργασία και να εργάζεται ο εργαζόμενο, αυτό πρέπει να νιώθει ασφαλή. Εξού και ερωτήσει μου. Τι πιστεύετε, η πρόταση αυτή θα μπορέσει να βγάλει τον κόσμο από την κρίζα αγορά εργασία, την κρίζα οικονομία, γιατί η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλιώ είναι στι σκανδιναβικέ χώρε, αλλιώς ε, στις ε, ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, κεντρικές. Είναι όμως πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να δουλεύουν νόμιμα και να καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση και να νιώθουν ασφαλείς. Άλλη ερώτηση. Είπατε ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά βάση γνωρίζει γιατί. Μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς πού μπορούν να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να την προχωρήσουμε αυτή τη συμφωνία και να την πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νόμιζα ότι με είχατε ξεχάσει, γι' αυτό έκανα χειρονομίες πριν. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι για την πρωτοβουλία σας αυτή κυρία Επίτροπε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επισφαλείς θέσει εργασία. Αυτό είναι ο στόχος μας. Πρέπει να δούμε όμως και ποιε είναι οι συνέπειες των φιλελεύθερων νόμων που συσσωρεύονται εδώ και δεκάδε χρόνια. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την επισφαλή εργασία. Και αν το δείτε, εσείς πηγαίνετε αντίθετα στο ρεύμα. Εμένα δεν με ενοχλεί, εμένα μου αρέσει να πηγαίνει κανείς ανάποδα στο ρεύμα. Αν δει κανείς τι έχει γίνει στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από τους νόμους Άλταν αλλά όχι μόνο και πιο πριν, βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να μειώσουν το κόστος εργασίας, πλήττοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Πολύ χαζό και ανόητο. Κάθε κυβέρνηση με το που έπαιρνε την εξουσία αυτό προσπαθούσε να κάνει. Οπότε εγώ σας ενθαρρύνω να πάτε προς την κατάσταση που θέλετε. Θα δω που θα καταλήξει, αλλά η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή. Πρέπει επίσης να δούμε λίγο και τι συνηθίζεται στις διάφορες χώρες. Δηλαδή τι συνηθίζουν να κάνουν επιχειρήσεις. Εσείς δεν λέτε τίποτα, εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται προβλεψιμότητα ένας ε, ε, εργοδότης, αλλά κάποιοι δεν θέλουν απλώς γυαλιά, θέλουν κιάλια. Αυτό το βιομηχανία για παράδειγμα. Είναι ένας κλάδος που εδώ και δεκαετίες κάθε χρόνο έχει 30% περίπου εργαζόμενους που παίρνει από τα γραφεία βρέσος εργασίας. Ε, μη μου πείτε τώρα, δεν μπορεί να ξέρει μια τέτοια επιχείρηση αν σε ένα χρόνο θα χρειαστεί 30% τέτοιο προσωπικό αντί για μόνιμο. Λοιπόν, όλοι αυτοί τι έχουν, έχουν εβδομαδιαίες οι βάσεις εργασίας. Εσείς είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια εύλοχη διάρκεια είναι αυτοί εύλογοι. Το ξέρετε, τους λέμε την Παρασκευή το βράδυ κατά πόσο πρέπει να πάνε να δουλέψουν τη Δευτέρα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το διάστημα είναι εύλογο και αποδεκτό. Και μάλιστα αν δούμε τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στον Νότο κυρίως, αλλά και όχι μόνο, από το 2008, 80 ε, με 95% των συμβάσεων είναι περιορισμένου χρόνου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τις πρακτικές γιατί εντάξει καταλαβαίνω ένα εργοδότη μπορεί μερικέ φορέ να μην είναι σε θέση να προβλέψει αλλά μην μου πείτε ότι δεν μπορεί να προβλέψει το 30% του προσωπικού του Απλώ το κάνουν αυτό για να πιέσουν ακόμα περισσότερο του πιο ευάλωτου εργαζόμενου. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Σον Σάιμον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο. Στην πρόταση που δημοσιεύεται, μία από τις προτάσεις σας είναι ότι οι συμβάσεις 0 ωρών μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να δίνουν στον εργαζόμενο ένα ελάχιστο αριθμό ωρών. Αυτό θα είναι μια βελτίωση συμβασεις μηδέν ωρων μετα απο ενα διαστημα αλλά όχι αρκετή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις μηδενικών ωρών καθόλου. Στις παρατηρήσεις που κάνατε όμως, νομίζω ότι είπατε, έτσι το σημείωσα εγώ τουλάχιστον, ότι θα πρέπει πάντα να έχουν έναν ελάχιστο αριθμό ορών οι άνθρωποι. Το οποίο είναι πολύ σωστό. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Οι συμβάσει μηδενικών ορών αν εγγυάστε κάποιες ώρες, δεν είναι μηδενικές συμβάσεις, οπότε θα ήταν ένα βήμα. Δεν είμαι όμως σίγουρος τελικά. Αυτό εννοούσατε. Οπότε στο τέλος σας παρακαλώ διευκρινίστε το αυτό. Κατά πόσο πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση όπου όλες οι συμβάσεις θα είναι συμβάσεις που θα εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας στον εργαζόμενο. Ξέρουμε όλοι πώς ε, λειτουργούν αυτά. Και εντάξει, μπορεί να έχετε 100 ερωτήσεις, πώς θα τις απαντήσετε όλες, μερικές μόνο και σίγουρα θα μπείτε στον πειρασμό να αφήσετε απ' έξω τις πιο δύσκολες. Εν Εγώ όμως, ορίστε, ε, σας παρακαλώ, απαντήστε στη δικιά μου την ερώτηση, έτσι με έναν απλό τρόπο, με ένα ναι, με ένα όχι, γιατί είναι απλή. Μην την ε, παρακάμψετε παρακαλώ. Μίκαελ Τέλτσιν τώρα, που είναι νέο μέλος της Επιτροπής μας από τα συνδικάτα της Γερμανίας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα Με την νέα αυτή οδηγία ε, πιστεύω ότι θα σταματήσουν οι ανήθικες συμβάσεις μηδενικού χρόνου. Ε, αυτό άλλωστε αναφέρεται στο άρθρο 9 με τον περιορισμό όμως ε, ότι μπορεί να υπάρξει δουλειά ε, ε, ε, όπου να βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη ο εργαζόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω και άλλους ομιλητές στον κατάλογο, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις της κυρίας Τάισεν. Δεν θα ακούσουμε λοιπόν άλλες ερωτήσεις. Ε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Τάισεν. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στο Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και την εξαιρετική υπηρεσία διερμηνίας που διαθέτεται, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσπαθήσει κανείς να απαντήσει. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω σε όλες. Ε, αν δεν το κάνω είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος ή γιατί δεν καταφέρνω να σημειώσω όλες τις ερωτήσεις. Οπότε αν δεν σας απαντήσω παρακαλώ να επανέλθετε. Και σίγουρα θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε γιατί έχετε δικαίωμα στην απάντηση της ερώτησής σας. Λοιπόν, για την ευελιξία. Α, ναι, είχα πει ότι θα μιλάω λαδικά λέει η κυρία Τάισεν, Για την ευελιξία. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε την ευελιξία στην εργασία. Ναι, πράγματι. Η κυρία Ροντρίκες νομίζω πολύ σωστά είπε ποια είναι και η ουσία της πρότασής μας. Πράγματι, στόχος είναι να έχουμε μία ε, αγορά εργασίας που όσο και αν αλλάζουν οι μορφές να υπάρχει αρκετή ευελιξία ώστε κάθε σύμβαση εργασίας, είτε πρόκειται για νέες μορφές είτε όχι, να προσφέρει μια ελάχιστη προστασία. Αυτό. Και γιατί χρειαζόμαστε ελάχιστα δικαιώματα εκεί, γιατί θέλουμε σύγκληση στην Ευρώπη, έτσι, και στα κοινωνικά, θέλουμε περισσότερη ακόμα σύγκληση, άρα πρέπει να γίνει προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και επειδή πρέπει να φροντίσουμε να προσαρμόσουμε τους θεσμούς μας στην νέα ε, κατάσταση. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους πλατφόρμες, αυτοπασχολούμενους, είτε οποιαδήποτε άλλη νέα μορφή εργασίας, όπως και ονομάζεται αυτή, πρέπει να φροντίσουμε να καλύπτεται και αυτή και να προστατεύονται με δικαιώματα οι εργαζόμενοι όλων αυτών των μορφών εργασίας. Εμείς δεν θα πούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να μπει μέσα σε μία ε, σύμβαση όσον αφορά την ευελιξία. Αυτό θα το αποφασίσουν ε, οι κοινωνικοί εταίροι στις διάφορες χώρες, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να καλύπτονται ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι από ό,τι κατά το παρελθόν, να καλύπτονται και αυτοί που είναι εργαζόμενοι πλατφόρμες και αυτοί που έχουν ε, συμβάσεις χωρίς όρους κλπ θέλουμε να τους καλύψουμε όλους αυτούς. Γι' αυτό διαβρύνουμε το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Περισσότερο δηλαδή από ό,τι ήταν η οδηγία για τη γραπτή δήλωση. Ακριβώς επειδή στην οδηγία για τη γραπτή δήλωση μπορούσαν οι χώρες μέλη να αποκλείσουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και ακριβώς να παίζουν με αυτές τις διαφορές οι χώρες μεταξύ τους. Και έτσι εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονταν εκτός κάποιας κοινωνικής προστασίας και αυτό δεν το θέλουμε. Όσο περισσότερες τέτοιες μορφές ε, εργασίας ε, δημιουργούνται, τόσο περισσότεροι εργαζόμενοι θα αποκλείεται. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να υπάρχουν κάποιες κοινωνικές προστασίες που να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους. Δεν καταστρέφεται έτσι η ευελιξία. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη, για τη δημιουργία απασχόλησης, να υπάρχει ευελιξία. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε όσοι έχουν τέτοιες συμβάσεις να έχουν μία ελάχιστη προβλεψιμότητα για το πότε θα δουλέψουν και να υπάρχει κάποια διαφάνεια για να μπορούν να προγραμματίσουν και αυτή τη ζωή τους και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας τους. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Τώρα για την συμμόρφωση. Υπάρχουν κανόνες για την συμμόρφωση που προβλέπονται σε όλα τα κοινωνικά. Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Έχουμε την παραδοσιακή διατύπωση, τι θα γίνει αν δεν υπάρχει αυτή η συμμόρφωση, ότι πρέπει να ευθαγραμμίζονται οι εργοδότες κτλ. Και γι' αυτό μιλάμε και για τις πληροφορίες. Θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ακριβώς ώστε ο εργαζόμενος να ξέρει περί τίνος πρόκειται και να μπορεί έτσι και ο εργοδότης να διορθώσει τη στάση του. Θέλουμε μια θετική αντιμετώπιση αν λείπει πληροφορία που μιλάει για μερική απασχόληση, ε, τότε είναι υποχρεωμένο ο εργοδότης να το κάνει πλήρους απασχόλησης. Αν δεν αναφέρεται δοκιμαστική περίοδο στις πληροφορίες που δίνονται στον εργαζόμενο, τότε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δοκιμαστική περίοδος. Τελείωσε. Από την αρχή προσλαμβάνεται ο εργαζόμενος χωρίς δοκιμαστική περίοδο και προβλέπουμε και διάφορες άλλες διατάξεις για διάφορες περιπτώσεις. Πώς μπορεί να πάει στο δικαστήριο ο εργαζόμενος, πώς προστατεύεται από κακή μεταχείριση. Υπάρχουν ε, διάφοροι κανόνες που αναφέρονται στην, ε, ε, στην πρόταση που έχουν να κάνουν με τις αποδείξεις, πώς αποδεικνύονται κάποια πράγματα κλπ. Αν θα περιοριστεί η γκρίζα εργασία, δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται από τον εργοδότη, γιατί δεν έχουμε βρει έναν ορισμό που να μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή που να είναι τέλεια. Βασιζόμαστε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον ορισμό. Μέχρι τώρα η κοινωνική μας νομοθεσία λέει κάθε φορά τι είναι ο εργαζόμενος ή μένει στη χώρα μέλος να το ορίσει. Εδώ λέμε ότι τον ορισμό μας τον βασίζουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι το οποίο σε όλες τις χώρες μέλη ισχύει. Δεν θέλουμε κατακαιρματισμό γι' αυτό και δεν θέλουμε παρεκκλήσεις που επιτρέπονταν πριν από τις διάφορες χώρες. Θέλουμε ακριβώς αυτό να αποφύγουμε να υπάρχει εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο για να μην μένουν εργαζόμενοι χωρίς προστασία. Τώρα για τον εργαζόμενο αυτό τι σημαίνει. Όταν είναι αυτοπασχολούμενος γίνονται έλεγχοι από την επιθόρηση. Αυτό η επιθόρηση πρέπει να το δει. Κατά πόσο δηλαδή ο άνθρωπος αυτός τελικά ανταποκρίνεται στον ορισμό του εργαζόμενου ή όχι. Αν ανταποκρίνεται στον ορισμό του εργαζόμενου, πρέπει να πάει στην κατηγορία εργαζόμενο και όχι αυτοαπασχολούμενο. Αυτή νομίζω είναι μια πρόταση που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, αλλά δεν λέω ότι θα την καταργήσει πλήρως. Για να απαντήσω τώρα και στα σχόλια του κ. Καλβέ Σαμπών, του εισηγητή, ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Αυτό ισχύει για όλους βέβαια. Είπε ότι η πραγματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα και στα διάφορα μέρη του κόσμου. Ναι, εμείς στην Ευρώπη όμως έχουμε κάποιες προδιαγραφές που είναι κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Έχουμε μια κοινωνική οικονομία, θέλουμε ε, την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη να ε, προχωρούν παράλληλα, γι' αυτό και θέλουμε την προστασία των εργαζομένων. Αυτό κάνουμε εδώ. Ήταν και στην προηγούμενη οδηγία για την γραπτή δήλωση, αλλά αυτό θέλουμε εδώ να περιγράψουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι του 1991, έτσι. Δηλαδή πριν από έναν αιώνα θα λέγαμε μεταφορικά. Οπότε τώρα διαβρύνουμε το ε, πεδίο εφαρμογής, εξυγχρονίζουμε τι διατάξεις λέμε ότι η πληροφορήση πρέπει να δίνεται γραπτά από την πρώτη μέρα που ισχύει η σύμβαση και όχι δύο μήνες μετά όπως ίσχυε πριν και κάτι το οποίο είναι επίση εντελώς νέο είναι ότι προβλέπουμε ελάχιστα δικαιώματα τα οποία να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των συνδικάτων. Ξέρετε ότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρό μας. Τα σεβόμαστε πλήρως. Ζητήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, όπως προβλέπει και η συνθήκη, αλλά όπως είναι και η πεποίθησή μας, έτσι αλλιώς. Ζητήσαμε διαβούλευση. Μια πρώτη φορά και μια δεύτερη φορά, έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο της συνθήκης. Και τελικά καταλήξαμε μαζί τους ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Μαζί το αποφασίσαμε αυτό. Και στο Κέτεμπορκ, στην ε, διάσκεψη που είχαμε εκεί με τους κοινωνικούς ε, εταίρους, τους είπαμε, σας δίνουμε άλλον ένα μήνα. Είχε λήξει η προθεσμία, αλλά είπαμε, ωραία, έχετε άλλον ένα μήνα στη διάθεσή σας για να καταλήξετε σε συμφωνία. Εμείς αν το Δεκέμβριο έρχεται και μας πείτε έχουμε συμφωνία, ό,τι και να έχουμε κάνει θα το σταματήσουμε και θα σας ακούσουμε. Όμως τελικά δεν ε, έγινε αυτό. Και που διαφωνούν. Υπάρχουν δύο τμήματα στην πρόταση αυτή. Το ένα είναι η πληροφόρηση η οποία πρέπει να δίνεται στους ε, εργαζόμενους, πότε πρέπει να δίνεται και τι να περιλαμβάνει. Και το δεύτερο είναι τα ελάχιστα, οι ελάχιστες προδιαγραφές, το κανονιστικό. Για το πρώτο, νομίζω ότι λίγο πολύ μπορούν να συμφωνήσουν. Για το δεύτερο όμως, οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Και επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο δεύτερο, ε, κάποιοι είπανε ούτε για το πρώτο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Κάποιοι είπαν πρώτα να γίνουν διαπραγματεύσεις. Ναι, αλλά αυτό θα καθυστερούσε πάρα πολύ και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Θα τέλειωνε η θητεία μας και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τίποτα. Και θα ήταν πολύ κρίμα να μην έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση που επήγει. Αυτή ήταν η λογική λοιπόν που μας οδήγησε στη συνέχεια να κάνουμε εμείς την πρότασή μας. Τώρα, στην πρόταση αυτή όμως δίνουμε πολύ περιθώριο στους κοινωνικούς εταίρους. Κοιτάξτε το άρθρο 12 της πρότασης, το οποίο λέει ότι όποιες και αν είναι τελικά οι διατάξεις, τα ελάχιστα πρότυπα δηλαδή που ορίζονται, τα, οι χώρες μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αφήσουν την εφαρμογή ε, στα στους κοινωνικούς εταίρους. Αν οι κοινωνικοί εταίροι σε μια χώρα αποφασίσουν ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές και έρθουν σε ένα ισορροπημένο πακέτο, τότε μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει οτιδήποτε άλλο. Διάφορα άρθρα είναι ε, αφιερωμένα ε, τις συλλογικές συμβάσεις, τους κοινωνικούς εταίρους κτλ. Τώρα είναι οι μαθητευόμενοι, οι ε, interims, οι ασκούμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή. Έχουμε πολλές και διαφορετικές ρυθμίσεις στις διάφορες χώρες μέλη για τους μαθητευόμενους. Οι ορισμοί διαφέρουν κατά πόσο είναι εργαζόμενοι ή δεν είναι αυτοί. Είπαμε λοιπόν για τους μαθητευόμενους και λοιπά. Τι γίνεται με τους αυτοπασχολούμενους, ρωτήσατε. Και ο εθνικός νομοθέτης τι περιθώρια έχει για τον αυτοαπασχολούμενο. Είπαμε, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ελάχιστη προστασία σύμφωνα με αυτή την πρόταση. Όποιος δεν είναι εργαζόμενος δεν καλύπτεται από αυτή την πρόταση, άρα από τις εθνικές ρυθμίσεις οι αυτοαπασχολούμενοι. Η τεχνολογία, είπατε, πάει πιο γρήγορα από την νομοθεσία και γι' αυτό πρέπει να το προβλέψει η νομοθεσία. Εντάξει, εμείς ακριβώς έτσι προσπαθούμε να προχωρήσουμε ε, με την ρύθμιση αυτή, ώστε να αφήσουμε περιθώριο στις εξελίξεις. Αυτό που θέλουμε και το έχουμε πάντα πει, ότι ό,τι εξελίξεις και αν δούμε, παρακολουθούμε τι γίνεται και φροντίζουμε στη σχέση εργαζόμενου-εργοδότη οι εργαζόμενοι να έχουν πάντα την κατάλληλη προστασία. Και αυτό ακριβώς προβλέπουμε σε αυτή την πρόταση. Θα φροντίσουμε δηλαδή όλες αυτές οι ευέλικτες συμβάσεις να είναι έτσι ώστε να προσφέρεται προστασία στους εργαζόμενους ακόμα και αν εξελιχθούν οι μορφές εργασίας. Η κυρία Γιονγκέριους επίσης ρώτησε, αλλά νομίζω την κάλυψε. Τώρα, ρωτάτε, αν οι χώρες μέλη θέλουν, μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από ό,τι προσφέρει η πρόταση αυτή. Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως και μπορούν. Πάντα το λέγαμε αυτό. Το άρθρο 53 πάντα λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά είναι οι ελάχιστοι κανόνες αυτοί που εμείς θεσπίζουμε. Οι χώρες μέλη μπορούν πάντα να προσφέρουν περισσότερα, όχι λιγότερα. Κατά τα άλλα, για την Σουηδία. Σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε πολύ με τους κοινωνικούς ε, εταίρους. Υπάρχει το άρθρο 12, όπως σας είπα, που πιστεύουμε ότι αφήνει μεγάλο περιθώριο στους κοινωνικούς εταίρους. Και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα πολύ καλό σύστημα συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλο το περιθώριο που διαθέτουμε και μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα πρόκειται για ελάχιστη προστασία ε, ανθρώπων εργαζόμενων. Κάτι το οποίο χρειαζόταν Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν ο κοινωνικός πυλώνας είναι αρκετά ευρύς. Ε, να, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτήν την κοινωνική προστασία. Είπαμε ότι θέλουμε σύγκληση. Γι' αυτό σας παρακαλώ στηρίξτε αυτήν την πρόταση δεν πρέπει να τη στηρίζουν μόνο οι χώρες οι οποίες πρέπει να κάνουν ακόμα πολλέ προσπάθειες για να φτάσουν στις ελάχιστες προδιαγραφές, πρέπει να τη στηρίξουν και οι υπόλοιποι. Εμείς δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τους κοινωνικούς εταίρους να φέρουν σε πέρα στο ρόλο τους. Πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιδούς συναδέρφους σίγουρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο λόγος που αντιδρούν στην Σουηδία τη στιγμή που η πρόταση αυτή προβλέπει ελάχιστες προδιαγραφές και προς αυτή την κατεύθυνση θα ρίνει. Ε, για τον ορισμό των εργαζομένων, σε τι βοηθάει. Πάλι επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για την απόφαση του δικαστηρίου. Σε αυτό βασιστήκαμε. Προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή όχι για άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι για τίποτα άλλο που ήδη υπάρχει. Εδώ πέρα πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής της συγκεκριμένης. Εκεί χρησιμοποιούμε τον ορισμό αυτό. Τώρα κύριε Σάντερ και άλλοι ερώτησαν πώς θα επηρεαστούν πράγματα όπω έχει, όπως είναι η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση κτλ. Και πάλι ό,τι εδώ πέρα λέει το δικαστήριο και εμείς χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε μόνο για αυτή την οδηγία και πουθενά άλλου. Ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Όντως δεν είναι πάντα εύκολη σχέση εργαζόμενου και εργαδότη είναι διαφορετική στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης από ότι στην περίπτωση μιας μεγάλης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διάλογος. Υπάρχει αυτό στο κείμενο. Άμα το διαβάσετε θα βρείτε τις λεπτομέρειες. Δοκιμαστική περίοδος, έξι μήνες, λέει ο κύριος Μαν, είναι το ανώτατο. Αν πρέπει να είναι περισσότερο, αυτό θα το αποφασίσουν ε, οι κοινωνικοί εταίροι στις χώρες μέλη. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια λογική περίοδος. Έξι μήνες φτάνει, κατά τη γνώμη μας, για να αποφύγουμε καταχρήσεις με τεράστιες δοκιμαστικές περιόδους που ανανεώνονται κτλ. Η κυρία Ροτρίγκες επίσης ρώτησε τι γίνεται με την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση που λέει ο κοινωνικός πυλώνας. Εμείς θα έχουμε πρόταση για πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Στις 13 Μαρτίου προβλέπεται. Θα υπάρξουν συστάσεις και θα κάνει τη διαφορά Εκεί θα υπάρχει διαφορά για τους εργαζόμενους, μεταξύ εργαζόμενων και αυτοπασχολούμενων. Η αλήθεια είναι ότι τα συστήματα στις χώρες μέλη είναι εντελώ διαφορετικά για τους εργαζόμενους και για τους αυτοπασχολούμενους. Θα έχουμε πάντως συστάσεις με περισσότερες λεπτομέρειες. Με στόχο όσο γίνεται περισσότεροι από τους ανθρώπους που δουλεύουν επαμοιβή να καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να μπορεί κανείς να πάει από το ένα καθεστώς στο άλλο χωρίς να χάνει δικαιώματα. Και τους κοινωνικούς εταίρους θα είπαμε. Θα βοηθήσει να μειωθεί ο κόσμος που δουλεύει στη μαύρη. Ναι. Δεν θα υπάρχουν πια ψεύτο αυτό απασχολούμενοι. Είναι εργαζόμενος σύμφωνα με τον ορισμό, όπως είπαμε, αν δεν είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενος. Και αντίθετα στο ρεύμα λέτε. Μπορεί να πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα. Αλλά η γραμμή μας είναι ο κοινωνικός πυλώνας. Αντίθετα στο ρεύμα, όχι, εγώ νομίζω ότι πηγαίνουμε με το ρεύμα πρέπει να δούμε ποια είναι η εξέλιξη της πραγματικότητας στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Περισσότερη ευελιξία στις συμβάσεις, λιγότερο τυποποιημένες συμβάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι το ατυπικό δεν πρέπει να γίνει ο κανόνας, εντάξει. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν μια πιο σίγουρη δουλειά όσο περνάει ο χρόνος, σίγουρα. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με άτυπες μορφές εργασίας να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερες συμβάσει, πιο μόνιμες και ότι αυτό πρέπει να υπάρχει γραπτά. Δεν μπορεί να το απαιτήσει ο εργαζόμενος, αλλά θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να το συζητήσει ο εργαζόμενος και να μπορεί να έχει αυτή την ευκαιρία να αποκτήσει μια πιο μόνιμη σχέση εργασίας με τον εργοδότη του. Για τα γραφεία ευρέσεως εργασίας και τους εργαζόμενους που βρίσκουν έτσι δουλειά. Υπάρχει σχετική νομοθεσία και πρέπει να την τηρήσουμε. Πρέπει να φροντίσουμε να τηρείται βέβαια και για τις μηδενικών ορών συμβάσεις δεν τις απαγορεύουμε. Γιατί τι θα πούμε, μπορεί από μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, αλλά λέμε ότι όταν πρόκειται για 8 το μήνα, θα πρέπει να είναι. Δεν λέμε ότι οι μηδενικών ορών συμβάσεων ε, καταργούνται, αλλά ακόμα λέμε και όταν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, τα δικαιώματα ισχύουν για τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος για ανθρώπους που έχουν τέτοιες ε, συμβάσεις. Κοινωνική εταίρεια. είπαμε, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να ικανοποιήσω τους περισσότερους συναδέρφους με τις απαντήσεις μου. Φυσικά και συνεχίζεται η συζήτηση. Εύχομαι στον εισηγητή και τους κοιόδης ε, οι εισηγητές να απολαύσουν τη δουλειά τους, να ξέρουν ότι πρόκειται για πάνω από 2 και 3 εκατομμύρια ανθρώπους που θα υποφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά που δεν έχουν τώρα. Σίγουρα κάτι μπορεί να διορθωθεί ακόμα, πάντως εμείς Έχουμε πει ότι θέλουμε να καλύψουμε όλους τους εργαζόμενους με κοινωνικά δικαιώματα. Αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με ισορροπία, χωρίς να καταστρέψουμε την ευελιξία. Επιτρέπουμε ευέλικτες συμβάσεις, αλλά όλοι όσοι έχουν κάποια σύμβαση, όλοι να καλύπτονται από τα δικαιώματα αυτά. Σίγουρα πρέπει να συζητάμε πάντα πολύ με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργατών, με τους κοινωνικούς ε, εταίρους δηλαδή, και όλα να τα βάζουμε σε ισορροπία και να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση. Κάναμε μια πρόταση. Εμείς προφανώς και την βρίσκουμε ισορροπημένη. Εσείς κάποιοι από εσάς λέτε ότι δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε ελπίζοντας να καταλήξουμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάισεν ε, και ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτές τις τόσο λεπτομερείς ε, απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις που δεχτήκατε. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πάντα είστε διαθέσιμοι, πάντα έρχεστε ε, και ε, πάντα παρουσιάζετε μακροσκελώς τις προτάσεις. Και δεν ε, μπαίνετε σύμφωνας για να βγείτε αμέσως από την αίθουσα, να φύγετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν περνάτε λιγότερο χρόνο μαζί μας. Ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν εκπρόσωποι 28 διαφορετικών χωρών με διαφορές μεταξύ τους. Και ε, βεβαίω ε, οι βουλευτές ε, καλούνται να συζητήσουν, να λύσουν προβλήματα. Και εσείς στο δικό σας επίπεδο μπορείτε να βρείτε λύσεις και διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέψουν στα κράτη να <clears throat> προχωρήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις του και να βρουν λύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας σε αυτή την δύσκολη συζήτηση. Ευχαριστώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος, έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σημείον 10. Η ενδυνάμωση της ε, οικονομικής, ε, κοινωνικής ε, και χωροταξικής, γεωγραφικής συνοχής. Έχουμε τον εισηγητή μας. <laughs> Εγώ η ίδια ε, ε, It takes the view that... Η πολιτική συνοχή είναι η μεγαλύτερη και θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη επενδυτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. I'm on the wrong... We are on point. Α, όχι, δεν είμαστε στο 10, είμαστε στο 9, έκανα λάθος, έχουμε κι άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε πίσω, σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως. Πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι και να κινηθούμε αποτελεσματικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή σχετικά με το, την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το έτος 2018. Παρακαλώ κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ο κύριος Χριστόφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τις οποίες έχουν υποβάλει όσον αφορά την έκθεσή μου ε, ε, σχετικά με την ε, ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ε, χάρη σε όλους ε, εσάς, σε όλους τους συναδέλφους, ε, η εργασία θα είναι ισορροπημένη και θα αποτελέσει με τα σε ένα καλό σημείο εκκίνησης. 256 τροπολογίες έχουν υποβληθεί που σαφώς εμπλουτίζουν αυτήν την έκθεση. Βέβαια δυστυχώς ε, ε, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πλαίσια οπότε δεν θα μπορέσω να εντάξω μήκους τέλος πάντων της έκθεσης και της νομοδότησης και επομένως δεν θα μπορέσω να βάλω όλα τα στοιχεία τα οποία θέλω όσον αφορά την εκπαίδευση, όσον αφορά την έλλειψη αντιστοίχησης ανάμεσα στις δεξιότητες και τις ε, και τη ζήτηση. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ε, πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι και αμφιλεγόμενα ή διαφορετικά. Ε, εν πάση περιπτώσει εγώ εν είδη συμβιβασμού υποβάλλω 36 συμβιβαστικές τροπολογίες με τους χιώδεις να σας πω ότι είχαμε τέσσερις συνεδριάσεις, μάλιστα μία συνάντηση είχαμε σήμερα το μεσημέρι στη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος. και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, τις συμβιβαστικές τροπολογίες έτσι ώστε να επιτύχουμε ισορροπημένη, ε, έναν ισορροπημένο συμβιβασμό και θα μπορέσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά με την έννοια ότι θα μπορέσουμε να ε, συγκεράσουμε θέσεις οι οποίες πολύ συχνά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εμείς, ε, όπω σα είπα, κάναμε πολλέ ε, συναντήσει για το θέμα. Αυτό θα κάνουμε κι άλλες. Ε, αυτό που είναι σημαντικό σε σχέση με τούτο το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα μήνυμα το οποίο θα είναι ισχυρό, το οποίο θα είναι ενιαίο, αλλά και το οποίο θα είναι ορθολογικό όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόληση. Αυτά και ήμουν πολύ αποτελεσματικό νομίζω, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Χάβι Λόπες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ όπως και ο εισηγητής μας θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, την, τον εισηγητή αλλά και τους υπολείπους σκιώδης για την εργασία που κάναμε μέχρι τώρα. Ε, πραγματικά είμαστε πάντα σε πνεύμα πολύ καλής συνεργασίας και πνεύμα επικοδομητικό. Τώρα φτάνουμε στην ουσία του θέματος ε, και υπάρχουν βεβαίως κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ ουσιώδη ανάγκη να έχουμε αύξηση των ε, μισθών, ε, δείκτες ε, κοινωνικούς ε, για το εξάμεινο, ε, ελάχιστο εισόδημα, όπως είπε και το Κοινοβούλιο άλλωστε πρόσφατα, προστασία των παιδιών της παιδικής ζωής κλπ. Και τώρα συζητούμε αυτά τα θέματα ουσίας προσπαθώντας να εξεύρουμε κάποιες ε, ε, συμβιβαστικές ε, λύσεις και ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Δουλεύουμε με όπως σας είπα πνεύμα συνεργασίας και επικοδομητικό πνεύμα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ. Ουλρίκε Τρεμπέσιους. Απουσιάζει. Την αντικαθιστά κάποιος, όχι. Για να τούμ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κρίμα που συζητάμε την έκθεση του κυρίου Χέτμαν τώρα που έχουν ολοκληρωθεί εργασίε πάνω στο θέμα αυτό. Η έκθεση αυτή νομίζω ότι είναι καλογραμμένη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο εισηγητής και έχει βρει πολλές λογικές ε, συμβιβαστικές προτάσεις. Θα ήθελα όμως ε, να κάνω ε, λίγες παρατηρήσεις ε, στο όνομα της ομάδας ALDE για την έκθεση αυτή για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πετύχει τον στόχο απασχόλησης του 75%. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών ε, και θα πρέπει να βελτιωθούν τα ποσοστά ε, ανεργίας. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ανεργία, ναι, βλέπουμε την ανάγκη για μέτρα συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα ε, στις ανάγκες της κάθε χώρας. Ε, η μακροπρόθεσμη ανεργία μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους στη φτώχεια, ωστόσο ε, κάποιοι άνεργοι ε, εμποδίζονται από την γραφειοκρατία, για παράδειγμα όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις άτυπες μορφές κατάρτισης, πόσο μάλλον μεταξύ των μεταναστών. Θα πρέπει να καλύψουμε το κενό ανάμεσα στην στην ε, έλλειψη δεξιοτήτων ε, και στην ανεργία. Η ανεργία των νέων ε, βρίσκεται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, δυστυχώς, και η ανεργία... Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει ακόμα δυναμικό που δεν έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες, για παράδειγμα οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρίες ή οι πρόσφυγες. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα και ε, τα υψηλά επίπεδα φτώχειας ε, ε, εμποδίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Γι' αυτό είμαι ενθουσιώδης όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο. Αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε μια κοινή προσέγγιση για την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε μόνο για καινοτομία και ανάπτυξη της αγοράς εργασία χωρίς να μιλάμε για την επαρκή κοινωνική προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αποτελεί όμως ε, μια ε, αναλαμπή ελπίδα για πολλού Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Η Κωνσταντίν Κακούνεβα δεν είναι παρούσα. Η Πρόεδρο είναι εκτό μικροφώνου. Αντικαθιστά κάποιος την κυρία Κούνεβα, όχι. Η κυρία Σδανόκα. Ε, και εγώ αντικαθιστώ στο θέμα αυτό την ε, Jean Lambert που δεν είναι στο κοινοβούλιο σήμερα. Έχουν υποβληθεί συμβαστικές προτάσεις. Και για τους πράσινους ε, το σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ανάπτυξη δικτών που θα πρέπει να καλύπτουν και τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Δεύτερον, οι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ε, χρειαζόμαστε και οικονομικούς δείκτες που θα πρέπει να οδηγήσουν σε διορθωτικές ε, δράσεις σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανισορροπίες. Επίσης, ε, θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές στις χώρες για την ομαλή μετάβαση προς ε, την ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Τέταρτον, ε, πέρα από τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προωθήσει τις δημόσιες κοινωνικές επενδύσεις. Και τέλος, θα πρέπει να παραπέμπουμε σε συγκεκριμένες νομικές πράξεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με, τους πυλών, με τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Αυτά, αυτές είναι οι βασικές μας θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κανείς παρόν από το EFDD, όχι. ENF, κανείς. Δεν είχαμε κανέναν από την ΚΟΕ e που να εκπροσωπεί την κυρία Κούνεβα. There is no one left from uh, the Commission who wants to... Ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης είναι κανείς εδώ που να θέλει να προσθέσει κάτι. Κύριε Χέτμαν, ένα λεπτό για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ως συμπέρασμα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας υποσχεθώ ότι στο τελευταίο στάδιο θα προσπαθήσω να συμβιβάσω το νερό με τη φωτιά, να τα συνδυάσω. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία θα βρεθούμε. Δεν μπορώ όμως να υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω κιόλα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. 26 με 27 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και στις 2 Μαρ... στη δεύτερη του Μαρτίου την Ολομέλεια θα πάει στην Ολομέλεια. Και πάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και δαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 7η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι η συγκήτρια. Οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι η βασικότερη επενδυτική πολιτική στην Ευρώπη αυτή και πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα χρηματοδότησης όπως και στην προηγούμενη περίοδο. Επίσης, θεωρώ ότι το κοινωνικό ταμείο πρέπει να παραμείνει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για την ολοκλήρωση και για την ένταξη των εργαζόμενων στην αγορά εργασίας με μέτρα υπέρ της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της ε, ανεργίας και της φτώχειας. Επίσης υπογραμμίζω ότι όσο πιο γρήγορα γίνει η εφαρμογή και όσο πιο μικρό διάστημα ε, μεσολαβεί στην προγραμματική περίοδο, τόσο το καλύτερο. Και το Ταμείο για την Απασχόληση όντως δεν αρκεί, πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. Ωραία, δεν είναι τίποτα φοβερά Ναι, αυτά, αλλά στέλνουμε το μήνυμα, αν μη τι άλλο, ότι χρειάζεται ακόμα ένα υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων. Ο κύριος Πρίατο δεν είναι πια εδώ. Εσείς θα μιλήσετε για το ΕΛΚ. Ωραία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, κυρία Συγήτρια, για το σχέδιο εκθεσής σας που αποτελεί μια πολύ καλή βάση προβληματισμού και συζήτησης για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η πολιτική συνοχή. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε επικοδομητικές συνομιλίες για αυτό το θέμα. Η πολιτική συνοχή, όλοι το γνωρίζουμε, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο οικοδόμησης μιας αλληλέγγυας Ευρώπης που να βρίσκεται κοντά στους πολίτες της. Μια πολιτική από την οποία πρέπει να επωφελούνται όλες οι περιφέρειες και επιμένω στο όλες. Μάλιστα ως ε, αντιπρόεδρος ε, μιας τέτοιας περιφέρειας της Ile de France να ξέρετε ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι ρόλο παίζουν οι περιφέρειες στα πλαίσια της διαφορετικής πολιτικής και πώς συνεισφέρουν στην οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή. Και όλα αυτά είναι που πρέπει να μας κινητοποιήσουν ακόμα περισσότερο γιατί βρισκόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ιδιαίτερα δύσκολο, όπου καταλαβαίνουμε ότι επίγει να αντιστραφεί η τάση αυτή έλλειψης εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τους πολίτες της. Η συνοχή λοιπόν από μόνη της έτσι καλλιώς αποτελεί προστιθέμενη αξία. Επιπλέον όμως θέλω να αναφερθώ σε τρία προβλήματα που είναι λειτουργικά, μεθοδολογικά και που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Το πρώτο πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα όταν φτάνουμε στην εφαρμογή. Γιατί θέλουμε μια πολιτική συνοχής που να είναι απλή, αποτελεσματική και λιγότερο γραφειοκρατική. Το διοικητικό άχθος είναι πάρα πολύ μεγάλο σήμερα και πρέπει να υπάρχει μια αρχή αναλογικότητας όταν ελέγχονται τα προγράμματα ανάλογα με τα ποσά που διακυδεύονται. Δηλαδή οι απαιτήσει ελέγχου δεν πρέπει να είναι ίδιες για ένα σχέδιο 20.000 ή 200.000 ευρώ. Επίσης, το λέτε κι εσείς, πιο γρήγορα πρέπει να γίνεται η εφαρμογή, να υπάρχει απλούστευση, πραγματική απλούστευση. Όλοι έχουν να κερδίσουν αν εμπνευστούμε από κάποια πράγματα που ισχύουν ήδη για κάποια προγράμματα. Το H2020, το Horizon δηλαδή, ή άλλα για τα πανεπιστήμια. Φτάνει μία φορά online να συμπληρώσει κανείς το φάκελό του, παίρνει έναν αριθμό με νέα νούμερα δηλαδή και από εκεί και πέρα βάζοντας αυτά τα νέα νούμερα έχει πρόσβαση στο προφίλ του όπου διατηρούνται όλα τα διοικητικά του στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα αντίστοιχο σύστημα για την πολιτική συνοχής. Όλες οι υποψηφιότητες έτσι θα είναι παρούσες σε ένα πόρταλ. Ο κάθε υποψήφιος θα έχει ένα δικό του νούμερο και άρα μπορεί έτσι να έχει τα διοικητικά ε, στοιχεία. Ε, μπορεί κανείς να ενημερωθεί για αυτά τα στοιχεία, τα οποία θα έχουν ήδη καταγραφεί για ένα πρόγραμμα και μηχανικά ε, μπορούν τα στοιχεία αυτά να συμπληρώνονται και σε οποιαδήποτε άλλη αίτηση για άλλο πρόγραμμα που κάνει ο ίδιος υποψήφιος. Αποκεντρωμένο σύστημα λοιπόν. Δεύτερον, πρέπει να επιμείνουμε να λαμβάνονται ακόμα περισσότερο υπόψη οι διαφορές ενδοπεριφερειακά. Γιατί υπάρχουν ε, βέβαια πλούσιες ε, περιφέρειες που όμως έχουν μέσα πολλούς φτωχού και το αντίθετο. Ακριβώς στην περιφέρεια Ile de France, όπου είμαι εγώ αντιπρόεδρος, έχουμε πολύ πλούσιες πόλεις σε κάποια διαμερίσματα και άλλες πόλεις, το, το Δήμους μάλλον, το Σαντενή με τεράστια οικονομικά και κοινωνικά πρόβλημα, όπου τα μειονεκτήματα πολλαπλασιάζονται. Τέλος, συμπληρωματικός δείκτης για το ΕΠ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες που να ανταποκρίνονται περισσότερο στην, προ... στην πραγματικότητα σήμερα και βάσει αυτών να χορηγούνται κονδύλια. Εσείς, ήδη από τις πρώτες γραμμές, στην έκθεσή σας αναφέρεστε στην ανεργία, τα ψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων. Λοιπόν, ίσως τέτοια να είναι αυτά τα συμπληματικά κριτήρια, πέρα από το ΑΕΠ δηλαδή, ανακάτοικο, να χρησιμοποιούνται και τέτοια κριτήρια, ώστε η πολιτική συνοχής να λαμβάνει υπόψη της και αυτά τα κριτήρια στην χρηματοδότηση. Έπειτα περισσότερη απλούστευση, λιγότερη γραφειοκρατία, εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και τέλος πολιτική συνοχής που αναλαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και κοινωνικά κριτήρια. Κατά τη γνώμη μου όλα αυτά πρέπει να προσέξουμε και είμαι πεπισμένος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ ικανοποιητικά δηλαδή. Ευχαριστούμε, κύριε Ζήτια. Ο Κουτιέρης Πιέτο δεν είναι εδώ, η κυρία Γιονκέριος τότε. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ το Σέρτζιο. Και πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Πρόεδρο. για τη γνωμοδότησή της. Όντως αποτελεί ένα καλό σημείο κίνησης για τη συζήτησή μας. Για μας και για όσους θέλουν κοινωνικές πολιτικές, όντως πολλά μπορούμε να στηρίξουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό σημείο κίνησης όπως αυτή η γνωμοδότηση. Τώρα, δεν το ξέρω, μπορεί να ανησυχούμε υπερβολικά, αλλά ανησυχούμε μήπως γίνουν περικοπές στο Ταμείο Συνοχής μετά το Brexit και μετά τις ε, αλλαγές στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Και βέβαια δεν θα πω ότι η Ενεργειακή Ένωση, η Ενιαία Αγορά, η Ψηφιακή Ένωση είναι πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αν η κοινωνική συνοχή εξασφαλίζει τη σύγκληση προς τα πάνω και την ευημερία, επηρεάζει και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό και πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ όταν ετοιμάζουμε το πουδουπού μετά το 2020. Οι κοινωνικές επενδύσεις είναι ακόμα κάτω από τα επίπεδα πριν την κρίση και οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και πρέπει εμεί να τα θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη. Έχω εδώ μπροστά μου τη δήλωση της ομάδας μου κατά οποιασδήποτε προσπάθειας περιορισμού της φιλοδοξίας που έχουμε εμείς για την πολιτική συνοχής. Την έχετε. Και θέλω να κάνω και κάποιες δηλώσεις για το πώς η πολιτική συνοχή και αυτή η σύγκληση προς τα πάνω μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στα πλαίσια του Πουδουπού. Στις συζητήσεις λοιπόν τις σχετικές θέλουμε να ζητήσουμε προβληματισμό γύρω από την πολιτική συνοχής και το πόσο αποτελεσματική είναι υπέρ της κοινωνικής πρόοδου. Μπορούμε να πούμε ότι δεν τα καταφέραμε να πετύχουμε κατά το παρελθόν αυτή την κοινωνική σύγκληση προς τα πάνω. Παρά τις έντονες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμίσει με τους κοινωνικούς στόχους την πολιτική συνοχής. παρόλα αυτά παραμένουν οικονομικές και κοινωνικές διαφορές ανά την Ευρώπη. Και με την κρίση επιδεινώθηκε η κατάσταση. Στη γνωμοδότηση αυτή λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε νέους δείκτες για να μετρηθεί αυτή η κοινωνική σύγκληση έναν δείχτη κοινωνικής πρόοδου, π.χ. που να δείχνει ότι με ψηλό ΕΠΕ περιφέρειες δεν είναι απαραίτητα αυτές που έχουν και τις καλύτερες επιδόσεις στην κοινωνική πρόοδο. Ένα τέτοιο δείκτης κοινωνικής πρόοδου θα πρέπει να μπορεί να μετράει την πολυδιάστατη κοινωνική πρόοδο, ζητώντα από τις περιφέρειες να εντοπίζουν τις κύριες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους. Θα ήθελα να δείτε πώς μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτές τις ιδέες, πώς μπορούμε να μετρήσουμε δηλαδή την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Για ένα συντάντσικα τώρα, από το ECR. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την δήλωσή σας για τη συνοχή. Η χώρα μου, η Σλοβακία, μπορεί να ε, προσπαθήσει να πετύχει καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους πολίτες της και με βάση αυτές τις αρχές. Ωστόσο, οι πολίτες ε, δεν βλέπουν αρκετά τις θετικές πλευρές. Πιστεύουν μάλλον ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά οι διαθέσιμοι πόροι. Δεν μπορούμε όμως να κατηγορούμε γι' αυτό την πολιτική συνοχής. Ε, τα προβλήματα ε, υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αν κάτι δεν λειτουργεί καλά, εάν δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα πετύχουμε. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις ακούστηκαν και συμφωνώ με αυτές. Καταρχάς, αποδοτικότητα, επίτευξη αυτών αποτελεσμάτων και δεύτερον, να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες και τα προσόντα των νέων. Στου νέου βρίσκουμε πολύ δυναμικό και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Οι προτάσει μου, οι τροπολογίε μου θα επικεντρωθούν σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο σε εκπρόσωπο της Άλντε. Όχι. Δεν είναι κανείς παρόν. Όχι. Γκουε NGL. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για, οικονομική, για ε, πολιτική συνοχής ε, χωρίς να συνδυάσουμε αυτήν την πολιτική, μάλλον την έλλειψη πολιτικής συνοχής ε, και να τη συνδυάσουμε με την πολιτική για την ενιαία αγορά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Τα τελευταία χρόνια η πολιτική λιτότητας <clears throat> είχε πολλές ε, επιπτώσεις ε, που επιβάρυναν ε, την κατάσταση. Δεν προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε την συνοχή. Αντιθέτως είδαμε ότι η φτώχεια, οι ανισορροπίες έχουν ενταθεί. Και πιστεύουμε ότι οι πολιτικές συνοχής που πρέπει πραγματικά να υλοποιηθούν, πιστεύω λέω ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται ε, στις ε, στρατηγικές αποφάσεις ε, και των κρατών μελών, δηλαδή χωρίς προϋποθέσεις και αιρεσιμότητες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κάθε χώρας λέω ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε την πραγματική συνοχή και σε εδαφικό επίπεδο εάν οι πολιτικές αυτές δεν συνδέονται με δημόσιες πολιτικές σε στρατηγικούς τομείς ε, χωρίς υποστήριξη των παραγωγικών κλάδων χωρίς ε, μείωση των ε, διαρθρωτικών εξαρτήσεων των χωρών κτλ. Και επίσης πιστεύουμε ότι μια πραγματική πολιτική συνοχή θα πρέπει να περνάει από την ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και ο τελευταίος προϋπολογισμός για μία ακόμα φορά ε, είναι μειωμένος στον ε, τομέα που μας απασχολεί. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να ενισχύσει την συνοχή θα έπρεπε να έχει διπλασιαστεί έτσι ώστε η δημοσιονομική ικανότητα να είναι σοβαρή. Ε, και ε, θα έπρεπε να λαμβάνει και υπόψη ε, και το ΑΕΠ των χωρών. Ε, πολιτική λοιπόν διαρθρωτική, πολιτική επενδύσεων κλπ. Ε, εδώ θέλω να σημειώσω ε, και την από επιτάχυνση κατά κάποιο τρόπο την διαρκή μείωση της έντασης όσον αφορά θέματα όπως είναι το κλείσιμο των συνόρων, τα λιγότερα κονδύλια κτλ. Αυτά όλα εμείς δεν μπορούμε να τα προσυπογράψουμε στα πλαίσια της ε, ενίσχυσης των προγραμμάτων, της ε, βελτίωσης των προγραμμάτων ενίσχυσης ε, της συνοχής, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν άλλωστε και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλο μέλος εδώ. Η FTD, η Λάουρα είναι εδώ, όχι. ναι, αλλά δεν θέλει να πει κάτι. Ζωέλ Μελάν. Κύριε Μαρτάν, θέλετε να πείτε κάτι. Έχουμε χρόνο για να δώσουμε τον λόγο στην Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν είμαι και σίγουρη, λέει η Πρόεδρος. Ίσως από τον κύριο Λουίς Ντίξ να ακούσουμε δύο λόγια την Κομισιόν. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, θα είμαι πολύ σύντομος. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε πολλά από τα σχόλια και τις συστάσεις ε, που βλέπουμε στην ε, έκθεση. Εδώ μιλάμε για απλούστευση, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν πολύ πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στα ε, κονδύλια. Και βεβαίως ε, άκουσα ε, την, ε, ε, το επιχείρημα για περισσότερους πόρους. Ναι και ο Επίτροπός μου το ίδιο θέλει και βεβαίως και θέλει και περισσότερους κοινωνικούς δείκτες. Επομένως πραγματικά λόγω του ότι δεν έχω και πολύ χρόνο θα περιοριστώ σε αυτά τα σχόλια. Πάρα πολύ ωραία. 27 Φεβρουαρίου λίγη η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών μόνο στα αγγλικά το μεσημέρι. Η 21-22 Μαρτίου θα συζητηθεί στην ΕΜΠΛΕ και ε, στην, Επιτροπή, στην Περιφερειακή Επιτροπή λίγο αργότερα. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσω το λόγο αμέσως στην εισηγήτρια ε, τη κυρία Γνιέσκα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι εδώ έχουμε διαδικασία βάσει του άρθρου 54 και επομένως μονάχα για τις αποκλειστικές αρμοδιότητες επιρροπής απασχόλησης μπορούμε να ε, μιλήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση όλων στην αγορά εργασίας εξαρτάται από την γενικότερη κατάσταση στην αγορά εργασίας και την οικονομία λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την προετοιμασία ε, και τις ε, δεξιότητες ε, του ατόμου και της εκπαίδευσης την οποία μπόρεσε να συσσωρεύσει στη διάρκεια της ζωής του. Και επομένως σπουδές και εργασία, αυτά είναι τα δύο στοιχεία του της γνωμοδότησης. Κοιτάξτε, η προετοιμασία των νέων έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό σκοπό της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ε, είναι ένα από τα στοιχεία, άρα η ποιότητα της εκπαίδευσης μας ενδιαφέρει. Ε, και ο έλεγχος ποιότητας εκπαίδευσης είναι και ένας, της απασχόλησης είναι και ένας από τους τρόπους ε, βάσει των οποίων μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης. Δεύτερο, ε, είναι πολύ προχωρημένη σε τεχνολογικό επίπεδο η αγορά εργασίας στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς ε, λόγω αυτής της μεγάλης ψηφιοποίησης ε, έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη για εξειδικευμένους, ιδιαίτερα καταρτισμένους ανθρώπους ενώ ε, η ζήτηση για λιγότερο προσοντούχους ε, ε, εργαζόμενους μειώνεται διαρκώς. Το σύστημα εκπαίδευσης προσπαθεί να αντιδράσει, προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό αυτό, ωστόσο είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτή η οποία προσελκύει το περισσότερο κόσμο. Και εδώ προκύπτει ο φαύλος κύκλος, γιατί έχουμε όλο και περισσότερους διπλωματούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ευκταίο, γιατί έχουμε πολλούς νέους ε, που μπορούν να λειτουργήσουν ε, καλά ε, γενικά αλλά όχι απαραίτητα στην σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε ότι πάνω από 20% των νέων Ευρωπαίων δεν έχουν δεν διαθέτουν βασικές ικανότητες όπως ας πούμε ε, η δυνατότητα να αναγνώσουν και να κατανοήσουν ένα κείμενο. Είναι ένα είδος αναλφαβητισμού δεύτερου επίπεδου. 20% των νέων έχουν ε, ικανότητες πολύ βασικές. Ακόμα και αυτοί που έχουν διπλώματα από, τις, από ανώτερες σπουδές, ε, από ΤΕΙ, από πανεπιστήμια, δεν έχουν αυτές τις βασικές ε, δεξιότητες. Και επομένως αναρωτιόμαστε, χρησιμεύει πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω μια ε, πρόταση ε, εξ ονόματος της ΕΜΠΛ που είναι η εξής. Δεν χρειαζόμαστε να βελτίωση ε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά τα benchmarks τα, τα οποία χρησιμοποιούμε θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την ποιότητα. Δηλαδή να έχουμε ε, περισσότερα ε, ποιοτικά ε, στοιχεία και παραμέτρους και όχι τόσο ποσοτικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε ενδεχομένως να καλύψουμε τα κενά του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί χρειαζόμαστε κάποιες ε, ε, ε, συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που τοποθετείται κάπου ανάμεσα στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Μονάχα τα τεχνικά λύκεια και οι τεχνικές σχολές είναι αυτές οι οποίες δίνουν κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αλλά οπωσδήποτε οι νέοι ε, πρέπει να ε, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους ε, και με άλλα στοιχεία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης και διασυνδέσεις πασαρέλες ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο και τον κόσμο της εργασίας όσον αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις είναι λίγες, φτάνουν αργά, ε, δεν αντιδρούμε δηλαδή αρκετά άμεσα και αρκετά ευέλικτα. Ε, σας ε, καλώ λοιπόν να σκεφτείτε λίγο αυτή την διασύνδεση ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο και τον κόσμο της εργασίας. Φλάβιο Ζανονάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για αυτό το προσχέδιο γνωμοδότησης. Ε, είμαι σκιώδης από τους, σκιώ... τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα υποβάλω κάποιες ε, πολύ στοχευμένες τροπολογίες, κυρίως με την πρόθεση να ενισχύσουμε κάποια στοιχεία και κάποιες παραγράφους. Υπάρχει μία φράση που με εξέπλησε εξέπληξε είναι του ε, Μπόκλι από τον ε, καθηγητή από το ε, Χάρβαρτ και λέει ότι εάν η εκπαίδευση κοστίζει πολύ δέστε πόσο θα κόστιζε η άγνοια. E Η επένδυση στην εκπαίδευση και την ε, κατάρτιση είναι θεμελιώδου σημασία για να προκύψει οικονομική ε, πρόοδο και επομένω πρέπει οπωσδήποτε να, να επενδύσουμε σε μια εκπαίδευση ε, εγγυημένη για όλου, υψηλή ποιότητα, σε ένα κοινό και αμοιβαία αναγνωρίσιμο πλαίσιο ε, στον πυλώνα, έχουμε τον πυλώνα τον κοινωνικό, ο οποίος ε, προέκυψε ε, πρόσφατα και εκεί προβλέπεται η εκπαίδευση, η μαθητεία, προβλέπεται η μαθητεία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση που όμως θα πρέπει να είναι ε, καλής ε, ποιότητος ε, έτσι ώστε να επιτρέψει στους νέους να συμμετάσχουν πλήρως και στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Εάν θέλουμε αυτός ο πυλώνας να παραμείνει μονάχα μια καλή πρόταση και μια καλή ιδέα τότε εντάξει διαφορετικά όμως θα πρέπει όλα τα στοιχεία τα οποία εκεί αναφέρονται θα πρέπει να εφαρμοστούν με τρόπο ουσιώδη θα πρέπει επίση να δούμε το θέμα της αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση γιατί από εκεί προκύπτουν τα προβλήματα του αποκλεισμού της περιθωριοποίησης ε, κτλ. θα πρέπει να παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία την εκπαίδευση και τη διασύνδεσή της ε, με την κοινωνία μια κοινωνία και μια αγορά εργασίας που βρίσκονται σε διαρκή ε, τροποποίηση και που αλλάζουν διαρκώς. θα πρέπει να προβλέψουμε Ευχαριστούμε επομένως μέσα από την εκπαίδευση και κάποιες εγκάρσιες ε, ικανότητες και κάποιες ε, ε, επιπλέον δεξιότητες. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που δεν είναι σαφές. Στο σημείο 6 του σχεδίου γνωμοδοτήσής σας, εκεί που αναφέρεστε σε νέες δεξιότητες τις οποίες πρέπει να περάσουμε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι λέτε εκεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν καλύτερη και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, μεταξύ των ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων και στις ε, μαθητείες και στα στάζ και σε οποιασδήποτε άλλες ανταλλαγές ε, <clears throat> θα πρέπει ε, να γίνονται λέω χωρίς κόστος ε, ε, ή εν πάση με πάρα πολύ μικρό κόστος. Περίπου 60% των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο παραμένουν χωρίς δουλειά και χωρίς οποιαδήποτε δραστηριότητα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ενεργούς πολίτες τους νέους. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τι προσπάθειε τους, να τι εντείνουν έτσι ώστε να ε, ξαναφέρουν ε, στην εκπαίδευση αυτά τα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει είτε το δημοτικό είτε και το γυμνάσιο θα πρέπει να ανοίξουν νέες, εργα... Ε, ε, ε, προϋποθέσεις και νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μέσα από νέα προσόντα. Να προβλεφθούν για τα... τους ανέργους, για τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, συγκεκριμένα προγράμματα. Κυρίως για την τελευταία κατηγορία πρόσφυγες και μετανάστες θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε την δυνατότητα να τους προσφέρουμε νέες δεξιότητες πολίτες νέες γνώσεις, νέες ικανότητες έτσι ώστε να ενταχθούν καλύτερα στην χώρα που τους φιλοξενεί. Επίσης θα πρέπει να ε, προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα και καταστάσεις για την ε, ε, εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να ενταχθούν. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια, ένα σύστημα αμοιβαίας αξιολόγησης και αναγνώρισης έτσι ώστε όλοι να μπορούν εντός της Ευρωπαϊκής να έχουν αναγνωρισμένο ορισμένα πτυχία. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητή, την εισηγήτρια, του κοιόδη κλπ. Ευχαριστώ, Άννα και δεν είναι παρόν. Τον αντικαθιστά κανεί όχι. Άλτε. Ε, δεν είναι παρόν η Ιωσένκο Εσελίμοβιτ, ούτε τον αντικαθιστά κάποιο, Ο Νεοκλής Ηλικιώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για το σχέδιο της νομοδότησης και για τη δουλειά που έχει επιτελέσει. Ε, από την πλευρά μας ως GUNGL έχουμε δυστυχώς ανησυχίες για το σχέδιο πρόταση νομοθέτηση που έρχεται μπροστά μας. Ως γενική αρχή εμείς θεωρούμε πως η εκπαίδευση πρέπει να, να παραμείνει ευθύνη του κράτους. Να είναι δημόσια και να είναι ανθρωποκεντρική εκπαίδευση. Και όταν λέμε ανθρωποκεντρική πάντοτε πρέπει να έρχεται στο νου μας ε, το τι είπε και έγραψε ο πατέρας της, ο φιλόσοφος της παιδείας ο Αριστοτέλης, ότι ο χρήσιμος άνθρωπος είναι ο άνθρωπο που συμμετέχει στα κοινά, ο ενεργό πολίτη. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε την εκπαίδευση. Ε, και να προσφέρει μια εκπαίδευση που θα προσφέρει ε, στι νέε γενιέ ομαλή πρόσβαση στον κόσμο τη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι η οργανωμένη κοινωνία, οι κοινωνικοί φορεί πρέπει να συζητούν με την πολιτεία τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών. Δεν πρέπει οι εκπαιδευτικέ πολιτικέ και ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να διαμορφώνονται από τι πολυεθνικέ εταιρείε για τις ανάγκες της δικής τους κερδοφορίας. Ε, θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια ε, εκπαίδευση ανθρωποκεντρική και όχι χρησιμοθυρική εκπαίδευση η οποία να υπηρετεί την αγορά. Θέλουμε μια εκπαίδευση που να υπηρετεί την κοινωνία. Είναι σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώ που η έκθεση επικεντρώνεται πάρα πολύ στην αντιστοιχεία δεξιοτήτων μεταξύ τη εκπαίδευση και τη αγορά εργασία. Αφήνει έξω προβλήματα όπω η όλο και περισσότερη δημιουργία επισφαλών εργασία, που θεσμοθετούν την επισφάλεια επικαλούμενη την εκπαίδευση και ε, οι πρακτικές ασκήσεις επιρετούν. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ψηφιοποίηση της εργασίας, διαμορφώνοντας το επιχείρημα επειδή η εργασία ψηφιοποιείται, υπάρχει αναντιστοιχεία των εργασιακών δεξιοτήτων, άρα δημιουργείται ανεργία. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε αυτό το επιχείρημα. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ ξεκάθαροι πω η ψηφιοποίηση τη εργασία δεν σημαίνει και απάλληφη επαγγελμάτων χαμηλών δεξιοτήτων. Σημαίνει σε πολλέ περιπτώσει τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων σε αυτά τα επαγγέλματα. Κατά συνέπεια, η εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων δεν σημαίνει και αυτόματα δημιουργία νέων ασφαλών και μόνιμων θέσεων εργασία. Αντίθετα, Ω Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρέπει να διασφαλίσουμε όπω η εργασία στην εποχή τη ψηφιοποίηση θα διασφαλίζει όλα τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Τέλο, σε μια κατανόψη μα περίεργη διατύπωση, στο σημείο 6, ε, λέει ότι δεν μπορούμε πλέον να σκεφτούμε με του όρου, δουλεία και θέση εργασία. Θεωρούμε πω η έκθεση δεν προωθεί με αυτήν την διατύπωση τη διασφάλιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα με τέτοιε ε, αναφορές προωθούμε την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Η ίδια η Επιτροπή μας θεωρεί ως την ψευδοπασχόληση και αυτόν καταγράφηκε σε πάρα πολλέ εκθέσεις ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο της εργασίας σήμερα και καταδίκασε αυτήν την ψευδοπασχόληση ε, πλήστες τόσες φορές. Η πρόθεση δίθεν εναλλακτικών μορφών απασχόληση πέραν τη εργασία ή τη δουλειά, δηλαδή μορφών τη προσφορά υπηρεσιών με ανάληψη ευθυνών από τον εργαζομένο, αναιρεί το δομικό στοιχείο τη ανάληψη τη κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου από τον εργοδότη του και από το κράτο. Εμεί ε, θέλουμε ξανά να ευχαριστήσουμε την ε, εισηγήτρια. Εμπολή ω ομάδα θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και θα καταθέσουμε ε, τροπολογίε που θα κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank ε, Ευχαριστώ πολύ, η Πράσινη Τέιραν και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, την συγγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι αποτελεί πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας να σας περιγράψω την κατεύθυνση προς την οποία ε, θα κινηθούν οι ε, τροπολογίες μας. Κι άλλοι αναφέρθηκαν ε, στην ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και ρομποτοποίηση. Εάν κοιτάξετε τις μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολύ διστάμενε απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας και νομίζω ότι στο σχέδιο έκθεση η γραμμή που ακολουθείτε είναι ότι με τις τάσει αυτές θα χρειαστεί να έχουμε διαφορετικού είδους εκπαιδευτικά συστήματα με το οποίο συμφωνώ, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να εξετάσουμε τι είδους βασικές δεξιότητες, τι βασικά προσόντα θα πρέπει να ε, έχει ο κόσμος για να μπορέσει να επιβιώσει σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει. Διότι ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν όλες οι μελέτες είναι ότι θα εμφανιστούν πολύ σύντομα νέες τάσεις για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμάζει το εκπαιδευτικό σύστημα τις μελλοντικές γενιές ε, σπουδαστών. Κάτι επίσης στο οποίο συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές είναι ότι ε, στην ανάλυση της κατάστασης σήμερα και όσον αφορά την ε, ανεργία γενικά αλλά ειδικά την ανεργία των νέων το θέμα αυτό συνδέεται πολύ με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, που οδηγούν στην υψηλή ανεργία και τα μέτρα λιτότητας των τελευταίων ετών ε, έχουν παίξει κάποιο ρόλο καθώς και το θέμα του πόσα χρήματα επενδύθηκαν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και κάτι ακόμα που θα θέλαμε να ενισχυθεί στην έκθεση αυτή είναι ο ρόλος ε, της διαβίου μάθησης, διότι όποια μελέτη και να κοιτάξετε ε, παρούσα, παρούσα είναι πάντα η αλλαγή στην αγορά εργασίας. Ε, η ιδέα ότι κάποιος στα 20 κάτι του θα κάνει την ίδια δουλειά μέχρι το τέλος της ζωής του δεν υπάρχει πια, δεν ισχύει πια. Συνήθως ε, κοιτάμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα υπάρχουν όμως ε, και άλλες μορφές μάθησης και απόκτησης προσόντος στο μέλλον και ε, θα πρέπει να αναφέρεται και αυτό στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λάουρα Ατζέα, EFTD. E Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε τη συνάδελφο Κουσλόφσκα για το προσχέδιο ε, γνωμοδότησης για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, τώρα βλέπουμε βεβαίως ότι η κοινωνία αλλάζει, περνάει από την βιομηχανική στη μεταβιομηχανική περίοδο. Μία περίοδο και μία εποχή με πολλά υλικά αγαθά ε, ε, που ε, πλέον δίνουν τη θέση τους όμως και σε άειλα αγαθά ψηφιοποίηση κλπ. Αυτό μας οδηγεί στο να αναρωτηθούμε ποιες θα πρέπει να είναι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και πώς μπορούμε να ε, δώσουμε μια νέα μορφή στην εκπαίδευση χωρίς όμως να την απογυμνώσουμε και χωρίς ε, να ε, την αφήσουμε καινή νοήματος. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με μέτρο και προσοχή γιατί ε, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογίες οι οποίες ε, θα εφαρμοστούν ε, και στις νέες και στη νέα αγορά εργασίας η ψηφιοποίηση γίνεται, λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον όπου οι αλλαγές πλέον γίνονται με ταχύτατο ρυθμό, ε, ε, με ρυθμό που πολλές ε, φορές αποσταθεροποιεί την κοινωνία μας τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούν σε αυτές τις ε, αλλαγές. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, θα πρέπει να ε, υπάρχει μια ομοιογένεια όσον αφορά τα προσόντα ε, και όσον αφορά τις δεξιότητες. Πάντως είναι απαραίτητο να έχουμε και μια άοκνη εργασία όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και την διαρροή ε, εγκεφάλων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την αποδυνάμωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου που διαπιστώνεται σε πολλές χώρες. Επίσης, η εγκατάλειψη, πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ έντονο, το οποίο έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο λόγω της κρίσης ε, που έχει ε, αυξηθεί και που έχει αυξήσει τις ε, ε, ανισορροπίες και τις αδικίες. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μονάχα αναλφαβητισμό όσον αφορά τα ψηφιακά. Έχουμε και μία αναζωπήρωση του αναλφαβητισμού με την πρώτη του έννοια. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε θα πρέπει να αντιδράσουμε και στις μεγάλες μειώσεις των κονδυλίων για την εκπαίδευση. Αυτή η τρομακτική τακτική μείωση των κονδυλίων, αυτή η γραμμική μείωση των κονδυλίων και των πόρων για την εκπαίδευση δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, πρέπει οπωσδήποτε και να προσαρμόσουμε και να εξυγχρονίσουμε και τα κτίρια των σχολείων και των πανεπιστημίων μας που καταραίουν αυτή τη στιγμή. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτά τα βασικά βήματα έτσι ώστε ε, η εκπαίδευση να μπορέσει να ακολουθήσει το βήμα και το ρυθμό των αλλαγών στην ε, κοινωνία. Θα πρέπει μέσα από φιλόξενες ε, εκπαιδευτικές δομές ε, τα, οι νέοι άνθρωποι να ε, αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για τις νέες μορφές εργασίας. Γιατί οι νέοι έχουν ε, απομακρυνθεί από την εκπαίδευση και δυστυχώς χάνεται αυτό το τεράστιο δυναμικό του διδακτικού προσωπικού ε, που έχουμε στις ε, χώρες μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν και να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να ξανασυνδέσουμε και τους διδάσκοντες στην διαδικασία αυτή. Τέλος, ε, η διασύνδεση ανάμεσα στο σχολείο, την εκπαίδευση και, το, και την ε, εργασία ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για ενδιάμεσες πασαρέλες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για μαθητείες, για στάζ που όμως δεν μπορεί να αποτελέσουν μορφή αδήλωτης εργασίας αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν μονάχα ένα μέσο μέσω του οποίου θα μπορέσουν να αποκτήσουν οι νέοι νέες δυνατότητες. Ε, να μπορέσουν μέσα από μαθητείες και μέσα από ε, ασκήσεις να αποκτήσουν νέες ε, δεξιότητες. Όχι όμως να δουλεύουν τζάμπα για πολυεθνικές εταιρείες, για μεγάλες εταιρείες οι οποίες θέλουν είτε τζάμπα τέλος πάντων είτε με πολύ χαμηλό κόστος να έχουν νέους εργαζόμενους. Uh, Ευχαριστούμε. Ε, κύριος Μαρτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια, σπάνιο από την πλευρά μας, για το εξαίρετο έργο της όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα στην Ευρώπη για να περιοριστεί η ανεργία. Και νομίζω ότι είναι πολύ πλήρης η έκθεσή σας, τόσο όσον αφορά την διάγνωση, όσον αφορά και τις συστάσεις. Εξυγχρονισμό, συνεργασία με την αγορά εργασία, εγκατάλειψη του σχολείου, ε, μαθητεία, δοκιμαστική περίοδος άσκηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ζήτηση δεξιοτήτων και από την άλλη μεριά το χαμηλό επίπεδο, όλοι το είπαμε, των νέων Ευρωπαίων. Ακόμα και όταν αυτοί έχουν διπλώματα πολλά. Εξάλλου, χαίρομαι, κυρία Συγήτρια, που επιτέλους για πρώτη φορά το δικό σας σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώνεται απλώς και μόνο στο στόχο του κειμένου, τον εξυγχρονισμό δηλαδή της εκπαίδευσης, χωρίς να έχετε συμπεριλάβει όπως γίνεται συνήθως τη συνήθις λέξη κλειδί, κυρία Πρόεδρε που οι Βρυξέλλες θέλουν να βάζουν μέσα σε όλες τις εκθέσεις τους. Μετανάστες, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλπ. κλπ, κλπ. Εσείς λοιπόν είχατε αυτή την καλή ιδέα να μείνετε πιστοί στο κείμενο και να μην μπερδέψετε το δικό σας μήνυμα και τις δικές σας προτάσεις με άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια. Πάντως, πολύ θα ήθελα να αναπτύξετε κάποιες ιδέες που είναι λίγο ασαφείς στο σχέδιό σας, την παρακολούθηση των διπλωματούχων. Με τι διαδικασία, ποιος θα το κάνει αυτό, ποιος οργανισμός, με τι κριτήρια ή ακόμα πώς θα ορίσουμε τις άτυπες ε, μαθητείες με τις επίσημες. Προτείνω να σας βοηθήσουμε, αν θέλετε. Θα σας βοηθήσουμε προτείνοντας τροπολογίες προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Κοβλόφσκα τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πραγματικά όλους σας για τις παρατηρήσεις σας. Συμφωνώ με αυτά που άκουσα. Συμφωνώ επίσης για το ότι η γνωμοδότηση αυτή μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο. Σε μια γνωμοδότηση ξέρετε ότι έχουμε μικρά περιθώρια, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλα κείμενα. Με τη βοήθεια τροπολογιών πάντως θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο σε διάφορα σημεία και να μην ξεχάσουμε έτσι τίποτα, να μην παραβλέψουμε τίποτα. Σίγουρα έχει και κοινωνικό στόχο η εκπαίδευση. Πρόκειται για την κοινωνική ένταξη ε, πρόκειται επίσης για την ε, διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία. Όλα αυτά που λέμε soft skills στα αγγλικά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ακριβώς πρόκειται για αυτές τις δεξιότητες, τις ήπιες, όπως τις λέμε, που δύσκολα τις παίρνει κανείς στο σχολείο. Συνήθως τις παίρνει εκτός σχολείου, γιατί το σχολείο, ακόμα και αν θέλαμε να κάνει κάτι διαφορετικό, το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές, όμως χαρακτηρίζεται από αδράνεια. Δηλαδή δεν προβλέπει, δεν προλαμβάνει τις αλλαγές, τις ακολουθεί. Οπότε πρέπει να βγει ο μαθητής από το σχολείο ή να εισάγουμε στο σχολείο τον εξωτερικό κόσμο για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η σύνδεση που λέτε. Ε, μιλάμε επίσης και για την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας. Ναι, αλλά μόνο 20 100 των σχολείων στην Ευρώπη διαθέτουν ψηφιακές υποδομές, υπολογιστές ή άλλες υποδομές για τους μαθητές τους. Οι περισσότεροι νέοι, δηλαδή οι πολίτες μας, δεν μαθαίνουν αρκετά τα ψηφιακά. Πώς λοιπόν θα προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας, πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αν δεν την έχουν μάθει στο σχολείο. Το σχολείο λοιπόν ε, σέρνει τα πόδια του, καθυστερεί, βρίσκεται πίσω, δεν ε, προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Άρα χρειάζεται να εισάγουμε αυτή την καινοτομία στα σχολεία, τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Και έρχομαι στο σημείο 6 για το οποίο με ρωτήσατε. Δεν είχα αρκετό χώρο, ε, γι' αυτό και δεν ανέπτυξε επαρκώ ίσω την ιδέα. Πάντω υπάρχουν πολλέ αναλύσει μέχρι τώρα που δείχνουν ότι υπάρχει δυναμισμό στην αγορά εργασία. Υπάρχουν νέα επαγγέλματα ή άλλα επαγγέλματα αλλάζουν και αλλάζουν συνεχώ. Η οργάνωση εργασία αλλάζει. Ο κόσμο είναι ασταθή, σε εξέλιξη. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξει η επιχειρηματολογία δεν πρέπει να επιχειρηματολογούμε βάση επαγγελμάτων, αλλά βάση κατηγοριών δεξιοτήτων. Αυτή είναι μια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής που ανταποκρίνεται σε αυτήν την αλλαγή επιχειρηματολογίας. Πρέπει να σκεφτόμαστε τις δεξιότητες και όχι τα επαγγέλματα. Πρόκειται για καθήκοντα, για αρμοδιότητε, για προσόντα, δεξιότητε που απαιτούνται για διάφορε θέσει απασχόληση. Και όταν τα κατέχουμε αυτά, μπορούμε να αλλάξουμε και δουλειά και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της θέσης απασχόλησης. Να αλλάξει το επιχείρημα λοιπόν, να αλλάξει η λογική και να ε, στοιχηματίζουμε περισσότερο σε μικρές διάρκεια καταρτήσεις με συγκεκριμένα προσόντα και διεξοτεχνίες. Το Harvard για παράδειγμα προσφέρει τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή προσφέρει κάποιες δεκάδες ώρες με μία ειδίκευση πολύ συγκεκριμένη και δίνει ένα πολύ ειδικό δίπλωμα. Αυτές οι μήνυ εκπαιδεύσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας με τέτοιου είδους διπλώματα και εφόσον συγκεντρώσουν πολλά τέτοια διπλώματα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Τέλος, για τον αναλφαβητισμό. Όντως πρόκειται για μεγάλη μάστιγα. Η έλλειψη βασικών προσόντων εμποδίζει τους νέους. Δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν να νιώσουν καν καλά στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν με τις τροπολογίες που υποβάλλω θα ζητήσω από τις χώρες μέλη να φροντίσει κανένα παιδί να μην φεύγει από το σχολείο χωρίς να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει μετά από 8 χρόνια από το σχολείο ένας μαθητής και να μην ξέρει να διαβάζει. Κάτι όμως που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να βγαίνει από το πανεπιστήμιο ένας νέος και να μην είναι σε θέση να γράψει και να διαβάσει. Κι όμως συμβαίνει αυτό μεγάλο ποσοστό των διπλωματούχων μας από τις ανώτατες σχολές δεν έχουν αυτές τις βασικές ικανότητες. Είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Αυτή η προθεσμία ε, υπολογή, υποβολής τροπολογιών είναι 28 Φεβρουαρίου στο 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε 21 και 22 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και 25 26 Απριλίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Πολιτισμού. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα, που είναι η έκθεση εφαρμογή τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πιμέντα Λόπε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η εκπόνηση μιας έκθεσης για ένα θέμα τέτοιο με τον περιορισμό που έχουμε όσον αφορά το μήκος της ε, καθιστά πολύ δύσκολο να καλύψουμε τις βασικές ιδέες μας. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση που θα έχουμε τώρα θα μας βοηθήσει ε, να ε, ε, διαμορφώσουμε καλύτερα το κείμενο και να παράσουμε έτσι κάποιες κατευθυντήρες γραμμές στην αρμόδια επί επιτροπή. Κάποιες παρατηρήσεις λοιπόν γνωρίζουμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε πολλά μέτωπα δύσκολα έχουν πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης, στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων, ε, στην ε, υγειονομική περίθαλψη, ε, σε υπηρεσίες που να αφορούν την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αθλητισμού. Επίσης ξέρουμε ότι η ανεργία των νέων είναι πολύ ανησυχητικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ανησυχητικά, ανησυχητικά συγγνώμη, τα στοιχεία. Έχουμε μια γενική ελαφρά, ε, ελαφρώς κατιούσα τάση, 18,7% ήταν η ανεργία των νέων ε, στα τέλη της περσινής χρονιάς. Ε, σε κάποιες χώρες το ποσοστό υπερεύει ακόμη και το 40%. Όπως και να έχει, Η μείωση της ανεργίας των νέων συνδέεται με ε, μορφές εργασίας που δεν μπορούμε να δεχτούμε, όπως είναι οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, ε, ε, θέσεις απασχόλησης, μερικής απασχόλησης κλπ. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τον αριθμό των νέων που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ε, ή φτωχοί και ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν λήψεις σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε την ε, οικονομική κρίση, Έχουμε τη διάβρωση των δημοσίων υπηρεσιών. Βλέπουμε όλο και περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης ε, με μη αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις, επισφαλείς εργασιακές σχέσεις κλπ. Υψηλό ποσοστό των νέων ε, βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης και δεν επενδύουμε επαρκώς στους νέους, στη νεολαία και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις με τη δημογραφική αλλαγή. Θα δούμε λοιπόν όλο και πιο πολλές επισφαλείς θέσεις εργασίας και αυτό με τη σειρά του θα ε, έχει αντίκτυπο στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. διότι δεν θα έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Λαμβάνουμε γνώση των συμπερασμάτων ε, της έκθεσης ε, για την ε, οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη που εκπώνησε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ο ILO. Οι 21 δισεκατομμύρια ευρώ χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα 2014 μέχρι το 2020 αν ε, είναι να πετύχει τους στόχους της. Ε, αλλά δεν διατίθεται τόσα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, ε, κάποιες πρωτοβουλίες για τους νέους για να προωθηθεί η απασχόληση. Έχουμε για παράδειγμα την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έχουμε την εγγύηση για την νεολαία. Ωστόσο, οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών είναι πολύ σημαντικές. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι μάλλον θλιβερή. Πρόσφατα συζητήσαμε σχετική έκθεση στην Ολομέλεια. όπου επισημάνθηκε ο περιορισμένος αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται. Δεν ε, επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα διότι δεν είναι επαρκώς ε, χρηματοδοτημένα. Έχουμε έκθεση για την προώθηση των αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, ε, την σημασία των συλλογικών συμβάσεων και την καταπολέμηση των επισφαλών εργασιακών σχέσεων. Την ανάγκη για δίκαιη αμοιβή. Πρέπει να παρέχουμε ε, καθολικές ποιοτικές υπηρεσίες και θα πρέπει να προωθήσουμε κοινωνικά προγράμματα τα οποία θα προωθήσουν την ε, ε, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη και την ευημερία των νέων. Χρειαζόμαστε επίσης προγράμματα και πρωτοβουλίες που να επικεντρώνονται στα προβλήματα αλλά και τις φιλοδοξίες των νέων. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την χρηματοδότηση για τις ε, πρωτοβουλίες για την νεολαία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι πολύ πιο καθολική και θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να μπορούν να φτάσουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Θα πρέπει δηλαδή να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων η χρηματοδότηση αυτή όμως δεν θα πρέπει να συμβάλλει έμεσα ή άμεσα σε μη αμοιβόμενε θέσεις πρακτικής άσκησης ή σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ούτε στην αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές θέσεις εργασίας ή με θέσεις πρακτικής άσκησης. Προσβλέπουμε στη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό και περιμένω να ακούσω τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πιμέντα Λόπες. Η Σοφία Ριμπέιρο απουσιάζει. Δεν την αντικαθιστά κανείς. Ήβα Πάνταρ. Παρακαλώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον ε, κύριο Λόπεσε για την ε, ε, γνωμοδότηση αυτή. Στη, επικεντρώνεται στην ανεργία των νέων που ακόμα βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα στα κράτη-μέλη. Επικεντρώνεται επίσης στην ανάγκη να επενδύσουμε στα δικαιώματα των νέων. Συμφωνώ ότι μια ενταξιακή πολιτική για την νεολαία συνδέεται και με την προώθηση των αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και θα πρέπει να βασιστούμε στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δημιουργικότητα καθώς και την ένταξη στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να τονιστούν περισσότερο κάποια θέματα στη γνωμοδότηση αυτή. Οι δυνατότητες πρακτικής ε, άσκησης, η ποιοτική πρακτική άσκηση, είναι πολύ σημαντικά θέματα. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εκμεταλλευτούμε τους νέους και να αντικαταστήσουμε ε, κανονικές θέσεις απασχόλησης με επισφαλείς ε, εργασιακές σχέσεις. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτά συμβόλαια, ε, να υπάρχει κοινωνική προστασία, αξιοπρεπής αμοιβή και αξιοπρεπείς ε, συνθήκες εργασίας. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης ε, θα πρέπει να οδηγούν σε ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης ε, και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να στηρίζουμε τις δομές των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να καλέσουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, να έρθουν σε επαφή με τους νέους, να τους επιτρέπουν περισσότερες δυνατότητες επιλογών και να τους βοηθήσουν να χτίσουν τη σταδιοδρομία τους. Έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε δει κάποια θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον τελικό μα στόχο. Ελπίζω η στρατηγική των νέων να εκπονηθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σεβάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Ε, τον εισηγητή, συγγνώμη, για τη γνωμοδότησή του. Θα κάνω ε, κάποια σχόλια. Βλέπω ότι στο, στο κείμενο γίνεται λόγος ε, περισσότερο για τη συμπερίληψη όχι τόσο για τις συλλογικέ συμβάσεις αλλά περισσότερο για την γενικότερη συμπερίληψη όλων των ανθρώπων. Οι νέοι άνθρωποι με ε, ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες. Ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν επίσης ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού, του, ε, τους. Επίσης ε, μπορούν, μπορούν να προωθηθούν διάφορες μορφές εθελοντικής μορφής εργασίας, μπορούν να δημιουργηθούν κέντρα στα οποία μπορούν οι νέοι να εργαστούν. Επίσης μπορούν νέοι στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας να, προσέχουν ηλικιωμένους κλπ. Οι τροπολογίες μου θα αφορούν ακριβώς αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, και ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ε, ε, προσχέδιο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω χωρίς να μακρηγορήσω είναι η γεγονός ότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εδώ μιλάμε για τα ε, για δικαιώματα των νέων. Δεν θέλουμε να δίνουμε φιλοδόρημα ή να, είμαστε, να δείχνουμε φιλευσπλαχνία προς τους νέους. Ε, οι νέοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να απαιτήσουν οι ίδιοι τα δικαιώματά τους ε, και να υλοποιηθούν τα δικαιώματα αυτά. Επίσης θα υπάρξει μία πρόταση ε, ε, σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι οι επενδύσεις ε, για τους νέους είναι επενδύσεις για το μέλλον και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές σε προγράμματα τα οποία αφορούν τους νέους και τη νεότητα, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό πρέπει να είναι ισχυρό σημείο της γνωμοδότησής μας. Τέλος οι οργανώσεις νέων. Οι οργανώσεις νέων συχνά ε, υποβιβάζονται με την έννοια ότι υποβιβάζεται ο ρόλος που παίζουν. Ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι οργανώσεις είναι ακριβώς αυτές μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να προωθήσουν τις ε, ιδέες τους, ε, μπορεί να ε, τους δώσουν τις πρώτες δυνατότητες έτσι ώστε να γίνουν πολύτιμα στελέχη της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που να ζητά το λόγο. τροπολογίες μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, ψηφοφορία 27-28 Μαρτίου, στην ε, ΚΑΛΤ 25-26 Απριλίου και στην Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που δεν τα παρατήσατε που μείνατε επί ώρες εδώ και ακούσατε όλες τις συζητήσεις και ευχαριστώ πολύ και τους καταπληκτικούς μας διερμηνείς. Λέει Πρόεδρος, την ευχαριστούμε. Γιατί και οι διερμηνείς ε, είναι εδώ πάντα, μας παραστέκονται στην προσπάθειά μας να συζητήσουμε και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Ευχαριστούμε.